So, dear colleagues, may we begin with the afternoon program. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινήσουμε το απογευματινό μας πρόγραμμα. Και θα ήθελα να καλωσορίσω την καθηγήτρια Γκίζελα Ρούλα, η οποία θα μας κάνει την παρουσίαση της ε, μελέτης για, ε, για το εμπορικό δίκαιο στα κράτη-μέλη είναι καθηγήτρια δικαιωμάτων του καταναλωτού και εμπορικών ζητημάτων και την έχουμε προσκαλέσει στο πλαίσιο της εκπόνησης έκθεσης πρωτοβουλίας για την ταχεία διεκπαιρέωση εμπορικών διαφορών. Έχετε το λόγο για περίπου 15 λεπτά και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από τους βουλευτές. Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να έρθω εδώ στο Κοινοβούλιο. Είχα έρθει και τον Ιούλιο για το θέμα των ε, εμπορικών διαφορών. Με μεγάλη χαρά έρχομαι να σας παρουσιάσω τις υπόλοιπες, ε, τα υπόλοιπα ευρήματα μου σε σχέση με την οικοδόμηση δυναμικού για την ε, αντιμετώπιση των εμπορικών διαφορών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Έχω τα εξή τμήματα στην ε, μελέτη. Καταρχάς ε, θα παρουσιάσω τις τα πιο σημαντικά ευρήματα και στη συνέχεια τις ε, συνέπειες που προκύπτουν από, από τα ευρήματα αυτά και στη συνέχεια τις συστάσεις που ελπίζω ότι θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της, του δυναμικού διευθέτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινήσω όμως με τα ευρήματα οι εμπορικές διαφορές αναπτύσσονται σε, μια πολύ σε ένα πολύ περίπλοκο οικονομικό ε, περιβάλλον γιατί αποτελούν ε, ένα μοσαϊκό διαφορετικών ε, κανόνων εθνικών, διεθνών και ευρωπαϊκών και έχουν ακόμα και προβλήματα ως προς την ασφάλεια δικαίου τα μέλη, τα μέρη μάλλον μια συμφωνίας όταν αναπτύσσουν διασυνοριακές συμβάσεις. Ε, και σε σχέση βέβαια με το δίκαιο που θα πρέπει να εφαρμοστεί. Έτσι λοιπόν πολύ συχνά ε, επιλέγουν ε, εφαρμοστέο δίκαιο, εφαρμοστέο στη σύμβασή τους και δικαιοδοσία που θα επιληφθεί της διαφοράς τους. Όταν το επιλέγουν αυτό λοιπόν πολύ συχνά επιλέγεται το αγγλικό δίκαιο και τα αγγλικά δικαστήρια. Αυτό μας δείχνουν οι εμπειρικές μελέτες, ότι πολύ συχνά το αγγλικό δίκαιο και τα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου επιλέγονται ως νομοθεσία και, δικαι... και δικαστήρια. Και πολύ συχνά οι επιλογές των μερών ε, ορίζονται από ποιοτικού παράγοντες, ποιότητα δηλαδή του αγγλικού εταιρικού δικαίου και ποιότητα των ε, δικαστηριών και δικαστών του Ρωμανού Βασιλείου. Είναι σαφές ότι η ικανότητα, το δυναμικό δηλαδή για την επίλυση εμπορικών διαφορών, όπως το αντιλαμβάνονται τουλάχιστον ε, τα μέρη σε μια εμπορική συμφωνία, ε, δεν έχει κατανόμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν ε, έχουμε μια σειρά από προβλήματα εντοπίσει από τις μελέτες μας. Καταρχάς ότι δεν έχουν όλοι οι έμποροι, όλες οι πλευρές, όλα τα μέρη σε μια εμπορική διαφορά τη δυνατότητα να καλύψουν το κόστος μιας τέτοιας διαφοράς ενώπιον των αγγλικών δικαστηρίων, τώρα μικρότερες επιχειρήσεις. Η προοπτική του Brexit βεβαίως ενισχύει τη δυσκολία καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο κατά πιθανότητα θα απολέσει την πρόσβασή του στον Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιοσύνη. Τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και η δικαιοδοσία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα έχει πλέον το πλεονέκτημα να ή το προνόμιο να διευθετούν δικαστικές διαφορές σε αστικά και εμπορικά ζητήματα επιπλέον η ε, δικαστές του Ρωμανού Βασιλείου δεν θα είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν, τουλάχιστον άμεσα υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν την, ε, τον κανονισμό γιώτα, ε, Βρυξέλλες ΙΑ και ενώ μέχρι τώρα οι, τα μέρη σε μια εμπορική σύμβαση ευχαριστώ επέλεγαν το Βρετανικό Φόρουμ, μπορεί να αρχίσουν να αναθεωρούν τις επιλογές τους αυτές. Ωστόσο, αν κοιτάξουμε το σύστημα διευθέτησης των αστικών διαφορών στα κράτη-μέλη, βλέπουμε ότι δεν ε, ανταποκρίνεται πάντα στις προσδοκίες των ε, μερών. Και είναι σαφές ότι υπάρχουν χώρες στις οποίες ε, μάλιστα τα μέρη μιας σύμβασης μπορεί να αποφεύγουν συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Δικαιοδοσία αυτό ισχύει για τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ιταλία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Ισπανία όπου οι ίδιοι οι εγχώροι έμποροι θεωρούν ότι είναι κακό το δικαιοδοτικό σύστημα και από το τελευταίο από τελευταία ε, το τελευταίο κατάλογο του World Justice Project, ε, αξιολόγηση δηλαδή της απονομής δικαιοσύνης, ε, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν ορισμένα κρατημέλη στα οποία δεν είναι ελκυστική η νομοθεσία και το δικαιοδοτικό σύστημα για τα μέρη μιας συμπορικής διαφοράς. Πράγμα το οποίο βεβαίως είναι πολύ δυσάρεστο, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και για το διασυνοριακό εμπόριο και για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς να μπορούν να εμπιστεύονται ε, τα μέρη, το δικαιοδοτικό σύστημα και να ξέρουν ότι μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια τη χώρα. Έτσι λοιπόν τίθεται το ερώτημα πώ μπορεί να βελτιωθεί, να ενισχυθεί περισσότερο το δυναμικό για απόδοση εμπορική δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα διατυπώσω μια σειρά από συστάσει λοιπόν με τη μελέτη μου. Η πρώτη έχει να κάνει με τη διαθέτηση διαφόρων στα κράτη-μέλη και την δυνατότητα εισαγωγή μια ταχεία διαδικασία για διασυνοριακέ εμπορικέ διαφορέ, αντίστοιχη με αυτή την οποία, η οποία έχει θεσπιστεί πριν από μερικά χρόνια για τις μικρής χαμηλής αξίας διαφορές. Η σύσταση λοιπόν σημειώνει ότι ένα από τα κύρια μελήματα των ε, μερών σε μια εμπορική συμφωνία στη διευθέτηση των διασυνοριακών διαφορών έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα και κυρίως την διάρκεια των ε, διαδικασιών. Υπάρχουν περιπτώσεις, παραδείγματι, όπου η ταχύτητα καταγράφεται ως ένας από τους πέντε κύριους λόγους για την επιλογή διαθέτησης μιας διαφοράς ε, με υπαγωγή στη δικαιοδοσία συγκεκριμένη χώρας. Και η ταχύτητα ή η απουσία ταχύτητα μπορεί να αποτελέσει ένα από του πέντε πρώτου λόγου για την αποφυγή υπαγωγή σε μια συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Πολύ συχνά βέβαια. Και είναι προφανές ότι είναι ελκυστικό ένα φόρουμ ε, μια ένωμη τάξη εφόσον μπορεί να προσφέρει ταχεία και αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνη. Δυστυχώ, ορισμένα κράτη-μέλη δεν πληρούν τι προδιαγραφέ αυτέ και από το EU Justice Corporate βλέπουμε πρόσφατα να καταγράφεται πω ε, οι αστικέ υποθέσει σε πολλά κράτη, αν όχι σε όλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κρατούν πολύ καιρό. Η παραδείγματι στην Ιταλία χρειάζονται περισσότερε από 500 μέρε για να δω, εκδώσει απόφαση ένα δικαστήριο πρωτοβάθμια σε εμπορικά ζητήματα. Στη Μάλτα, τη Σλοβακία, την Κροατία και την Ελλάδα χρειάζονται 400 ημέρε περίπου. Με δεδομένο αυτό, λοιπόν, μια ταχύτερη ευρωπαϊκή διαδικασία θα αποτελέσει ένα βήμα προόδου, γιατί θα εξασφαλίσει ότι σε κάθε κράτο μέλο θα υπάρχει δυνατότητα για μια ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία στη διάθεση των ε, μερών μια σύμβαση για τη διευθέτηση των διασυνοριακών του διαφορών. Ωστόσο, για διάφορου λόγου, δεν μπορεί να αποτελέσει πανάκια μια τέτοια ταχεία διαδικασία. Πρώτον, Οπωσδήποτε, βέβαια, σε ορισμένα κρατημέλη είναι χρονοβόρε αυτέ οι διαδικασίε, αλλά δεν έχουμε εμπειρικά δεδομένα που να μα εξηγούν του λόγου γι' αυτό. Εάν δεν υπάρχουν αρκετοί δικαστέ ή αν δεν υπάρχουν αρκετά καταρτισμένοι δικαστέ, μπορεί να επηρεαστεί η διάρκεια τη ε, δίκη, αλλά το ίδιο ισχύει και για την απουσία πόρων ή ε, ηλεκτρονικών υποδομών, πληροφορικέ δηλαδή. Δεύτερον, μπορεί όταν επιλέγουν ένα συγκεκριμένο φόρουμ ή ε, τα μέρη να το πράττουν για λόγους ταχύτητας, δεν είναι αυτός ο αποκλειστικός λόγος, γιατί υπάρχουν και άλλοι και πολύ πιο σημαντικοί λόγοι από ό,τι μας δίνουν ε, οι εμπειρικές μας μελέτες. Μια ταχύτερη λοιπόν διαδικασία θα μπορούσε απλώς να συμβάλλει στην ε, ταχύτερη στην εξασφάλιση καλύτερων αποτελεσμάτων σε ορισμένε περιπτώσεις, αλλά στις πιο περίπλοκες δεν είναι αυτό το μόνο κριτήριο. Τρίτον, μια καλύτερη διαδικασία δεν έχει κανένα νόημα εάν το δικαστήριο και οι δικαστέ δεν έχουν είτε αρμοδιότητα, είτε γνώσει είτε εμπειρία για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών εμπορικών διαφορών. Ε, στα αγγλικά δικαστήρια και ειδικά στο εμπορικό δικαστήριο του Λονδίνου, London Commercial Court, ε, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η προτίμηση όχι μόνο γιατί θεωρείται ότι είναι ταχεία και αποτελεσματική η απονομή δικαιοσύνη, αλλά και γιατί χαίρουν ιδιαίτερου σεβασμού οι δικαστές και θεωρείται ότι είναι ειδικοί στα θέματα του ε, εμπορικού δικαίου. Έτσι λοιπόν η εισαγωγή μια ε, ταχεία διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τι ασυνοριακέ και εμπορικέ διαφορέ δεν μπορεί παρά να είναι ένα πρώτο βήμα. Ένα δεύτερο βήμα, και το συνιστώ με τη μελέτη μου, με την έρευνά μου, θα ήταν η εγκαθίδρυση ειδικών δικαστηρίων εμποροδικίων για τι διασυνοριακέ εμπορικέ υποθέσει ε, στα κρατη και από τα κρατη Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζεται πως υπάρχει η εξειδίκευση και ότι αποτελεί αυτή το υπαριθμό ένα εργαλείο για την εξασφάλιση ποιότητας στις δικαστικές, ε, στην επίλυση εμπορικών διαφορών. Επί παραδείγματι, η Γερμανία έχει επιτυχημένα πειραματιστεί με εξειδικευμένα δικαστήρια στο πλαίσιο της δικαστικής συνδρομής και ειδικότερα στον τομέα των διεθνών ε, υιοθεσιών και μέτρων που αφορούν την προστασία των τέκνων των Σε μια... Ε, και αντίστοιχα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία έχουν συγκεντρώσει την εφαρμογή των... Ε, του κανονισμού για τις ε, διαφορές μικρής αξίας σε ένα συγκεκριμένο δικαστήριο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει παράδοση για υψηλή εξειδικευσή δικαστήρια στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία. Επίσης προβλέπεται με βάση τον κανονισμό Community Design, σχεδίου δηλαδή ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι, ότι απαιτείται να εγκαθιδρυθούν ειδικά δικαστήρια που ασχολούνται με το σήμα, το εμπορικό και το σχέδιο. Έτσι λοιπόν θα πρότεινα τουλάχιστον ε, κάθε κράτος μέλος να έχει ένα ειδικό δικαστήριο που θα ασχολείται με τις διασυνοριακές εμπορικές ε, διαφορές. Έτσι αυτό το δικαστήριο θα μπορούσε ταχύτατα να αναπτύξει και την εμπειρία και την εξειδίκευση γιατί θα επιφορτίζεται με, τις, ε, με ίδιου τύπου, με ομοίου τύπου υποθέσεις κυρίως. Και επιπλέον έτσι θα γνωρίζουν και τα μέρη ότι υπάρχει ένα ειδικευμένο δικαστήριο που θα μπορούσε να εκδικάσει την υπόθεσή τους. Θα ήθελα για το δικονομικό τμήμα να πω ότι θα πρέπει αυτά τα ειδικευμένα εμποροδικεία να εφαρμόσουν τις ταχείες διαδικασίες και μια πιο ευέλικτη για τις πιο περίπλοκες περιπτώσεις, ευέλικτη και ε, σχεδιασμένη ειδικά ε, διαδικασία για να καλυφθούν ε, οι ανάγκες ειδικέ των αλλοδαπών μερών ε, μερών προερχομένων από, τρίτο κράτος, από κράτος άλλο αυτού του δικαστηρίου θα πρέπει να γίνονται οι δίκες στα αγγλικά. Πιστεύω ότι αν υιοθετηθούν αυτές οι συστάσεις θα κερδίσει πολλά σε επίπεδο αποδοτικότητας και ε, ποιότητας των ε, εμπορικών δικών ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι υπάρχει ακόμη κάτι περισσότερο. Θα ήταν σκόπιμο ίσω να εγκαθιδρυθεί ένα διεθνέ δικαστήριο για την διευθέτηση των διασυνοριακών εμπορικών διαφορών, ένα ευρωπαϊκό εμποροδικείο, το οποίο θα ε, λειτουργούσε συμπληρωματικά προς τα δικαστήρια των κρατών μελών και έτσι θα εξασφάλιζε μία πρόσθετη και διεθνή δυνατότητα, μια διεθνή δικαιοδοσία για τη διευθέτηση των διασυνοριακών διαφορών με σημαντικά πλεονεκτήματα, ε, παραδείγματι και καταρχάς θα αποτελεί ένα πραγματικά διεθνέ δικαστήριο και ω εκ τούτου θα μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα αυτό το ευρωπαϊκό εμποροδικαίο στι ανάγκε των εμπορικών μερών, των ε, συμβαλλωμένων μερών, από ότι εθνικά δικαστήρια που ανήκουν μόνο στο υφιστα... στην εφιστάμενη τάξη, εθνική τάξη Και επίση θα μπορούσε να έχει περισσότερη εμπειρία, ουδετερότητα για την διευθέτηση, για την ε, κρίση διεθνών διαφορών. Θα μπορούσε ως ένα διεθνές διαιτητικό δικαστήριο, παραδείγματι, να ε, ε, έχει να, στους κόλπους του δικαστές εξειδικευμένους και έμπειρους στο εμπορικό δίκαιο από διάφορα κράτη-μέλη. Θα μπορούσε έτσι να συλλέξει την εμπειρία για τη διευθέτηση των διεθνών διαφορών. Και επιπλέον θα μπορούσε να προσφέρει πολύ περισσότερα και αποδοτικά αποτελέσματα για, τις, ε, ε, για τους αντιδίκους από, ένα εθνικό ευρώ, ε, από ένα εθνικό εμποροδικείο. Ταυτόχρονα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ένα τέτοιο ευρωπαϊκό εμποροδικείο θα μπορούσε και ξεπερνώντας τα όρια της απλής διευθέτησης των ευρωπαϊκών διαφορών να επομίζεται και τη διευθέτηση, την κρίση διεθνών εμπορικών διαφορών πολύ πιο αποτελεσματικά και πιστικά, όπως έχουμε δει ότι τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρει διαφορές που έχουν να κάνουν παραδείγματι με την Κίνα ή τη Σιγκαπούρη. Θα μπορούσε δηλαδή να αποτελέσει ένα ελκυστικό παγκόσμιο φόρουμ, ένα τέτοιο ευρωπαϊκό εμποροδικαίο για τη διευθέτηση διεθνών ε, διαφορών. Έτσι λοιπόν, θα πρότεινα τρία μέτρα συνολικά για την βελτίωση της ικανότητας κρίσης εμπορικών διαφορών. Πρώτον, εισαγωγή ταχείας διαδικασίας για τις διασυνοριακές διαφορές που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε επίπεδο ε, δικαστηρίων των κρατών μελών. Δεύτερον, εγκαθίδρυση ειδικευμένων εμποροδικαίων ε, εξειδικευμένων στον τομέα αυτό. Και τρίτον, ε, θέσπιση ενός ευρωπαϊκού εμποροδικείου. Επιπλέον, θα πρότεινα την ε, υιοθέτηση μια σειρά επιπλέον μέτρων που θα έχουν να κάνουν με την επιλογή της ένομης ε, τάξης, την κατάρτιση των δικαστών, την πρόσβαση στο αλλοδαπό δίκαιο, αλλά και την ε, νομική κατάρτιση. Για λόγους χρόνου δεν μπορώ να τα εκθέσω αυτά αναλυτικά, αλλά στα η γραπτή μας παρέμβαση μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες και πολύ ευχαριστούμε τη συζήτηση. Αν έχετε ερωτήσεις, να δώσω απαντήσεις. Θα ήθελα λοιπόν καταλήγοντας να επισημάνω πώς πιστεύω πως το προτινόμενο αυτό σύνολο μέτρων, εάν εφαρμοστεί, θα βοηθήσει στην βελτίωση της λογικής ε, ικανότητας απόδοσης δικαιοσύνης στο εμπορικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εξασφαλίσει πρόσβαση για τους ε, αντιδίκους εμπορικών διαφορών σε δικαστήρια υψηλής ποιότητας και σε διαδικασίες σε κάθε κράτος μέλος ανεξαρτήτως του μεγέθους ή του πόρου, των πόρων που έχουν στη διάθεσή τους. Επίσης θα μπορέσει να εξασφαλίσει ότι θα, θα γίνεται η επιβολή των ε, ε, αποφάσεων και η διεκδίκηση των απαιτήσεων πέραν των σύνορων ανεξαρτήτως της προελεύσεως των συμβαλωμένων. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να αποτελέσει έναν ελκυστικό πόλο για τη διευθέτηση και κρίση διεθνών εμπορικών διαφορών. Θα γίνει δηλαδή πιο ελκυστική ως χώρος που μπορεί κανείς να αναπτύξει τις εμπορικές του συναλλαγές. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Τώρα υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρία ε, για τους βουλευτές να θέσουν ερωτήσεις. Ο κύριος Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την ομιλήτρια. Μας έκανε πάρα πολλές συγκεκριμένες προτάσεις και ακριβείς. Είναι σπάνιο ένας ομιλητής σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να κάνει τόσο πλήρες προτάσεις. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτά που είπατε, δηλαδή αυτά που προτείνετε για να βελτιωθεί ένας διασυνοριακός ε, μηχανισμός εμπορικών ε, διαφορών στην Ευρώπη. Και πραγματικά χτίσατε και ένα suspense με τις προτάσεις σας. Με την πρώτη πρόταση δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή ότι ε, θα πρέπει τα εθνικά δικαστήρια να διεκπεραιώνουν ταχύτερα τις υποθέσεις 400 μέρες στην Ελλάδα, 500 μέρες στην Ιταλία, έχετε δίκιο. Δεν υπάρχει λοιπόν κριτική σε αυτό. Η δεύτερη πρόταση είναι ήδη κάπω ε, πιο δύσκολο να τεθεί σε εφαρμογή, γιατί προτείνεται να θεσπιστεί ένα ειδικό δικαστήριο σε κάθε κράτο μέλο για τι δυσυνοριακέ εμπορικέ διαφορέ. Και προφανώ μπορούμε να αρχίσουμε εδώ να αμφιβάλλουμε, γιατί κάθε φορά που έχουμε μια κάπως δύσκολη διαφορά, τίνουμε να στρεφόμαστε προς ένα ειδικό δικαστήριο. Όμως ε, αυτό ε, μου, κάνει, με, μου προκαλεί φόβο, γιατί διαφορετικά η εθνική δικαιοσύνη ε, ουσιαστικά θα κατηγορηματιστεί σε πολλά ειδικά δικαστήρια. Και τι θα μείνει για τα κοινά δικαστήρια του κοινού δικαίου. Έτσι λοιπόν, ε, θα θα πρέπει να έχουμε ένα δικαστήριο ευρείας αρμοδιότητας και φαντάζομαι ότι έχετε και ένα εναλλακτικό σχέδιο, γιατί νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να έχουμε ειδικά τμήματα. Νομίζω ότι θα δυσκολευτείτε να πείσετε τα κράτη να προσανατολιστούν προς τη λύση αυτή. Κατάλαβα νομίζω ότι είπατε ότι να υπάρχει μια διαδικασία στα αγγλικά σε αυτά τα δικαστήρια. Νομίζω ότι αυτό θα έθετε συνταγματικά προβλήματα σε κάποια κράτη, κυρίως στη Γαλλία όπου ακριβώς ορίζεται ότι τα γαλλικά είναι η γλώσσα της δικαιοσύνης. Και κλείνω με την πρότασή σας, την τελική, να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δικαστήριο. Εδώ δεν σας παρακολουθώ πολύ καλά, θα ήθελα μια διευκρίνηση. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό το εμπορικό δικαστήριο δεν θα αντικαθιστούσε τα ειδικά εθνικά δικαστήρια, αλλά θα ήταν κάτι πρόσθετο, ε, συμπληρωματικό. Πώς λοιπόν θα διαρθρωνόταν ε, η αρμοδιότητα αυτού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με τα ειδικά εθνικά δικαστήρια. Πρώτη ερώτηση ήταν αυτή, δεύτερη ερώτηση. Είδα στον πίνακα μία πληροφορία που δεν αναπτύξετε και με ενδιαφέρει πολύ. Έλεγε επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου, choice of law στα αγγλικά. Θα ήθελα να μου πείτε σε τι συνίσταται αυτό. Τι εννοείτε με αυτή την ε, επιλογή του εφαρμοστείου δικαίου. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ε, πάντως ήταν συναρπαστική η παρουσίασή σας. Κύριε Κάφμαν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο σχεδόν συζητητής κύριος Κονφεράτη ζητά συγγνώμη γιατί δεν μπορεί να είναι σήμερα στις Βρυξέλλες και μου ζήτησε λοιπόν να μιλήσω εξ ονόματός του. Του έτυχε κάτι απρόπτο. Θα ήθελα λοιπόν ο κύριος Κονφεράτη να σας ευχαριστήσει θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη σας. Και εξ ονόματο του κύριου Κομφεράτη θα ήθελα να μεταφέρω κάποιες ε, ερωτήσεις ε, για την διαπραγματευτική ικανότητα των μερών. Στην ε, αρχή της μελέτης είπατε ότι σε περιπτώσεις εμπορικών διαφορών οι δύο, οι δύο αντίδικοι βρίσκονται σε ίση θέση. Είναι ίση. Όμως θα μπορούσαν να υπάρχουν ανισότητες, για παράδειγμα, στην περίπτωση που ένας αντίδικος ε, χρήζει προστασίας. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες ε, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και ε, υστερούν σε διαπραγματευτική ικανότητα σε σχέση με τις μεγάλες πολυεθνικές. Και μάλιστα όταν μιλάμε για πολύ μικρές επιχειρήσεις, η διαφορά είναι τεράστια. Αυτή είναι η σημαντικότερη ερώτηση του κυρίου Κονφεράτη λοιπόν. Τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ε, άσχημη θέση, τη μειονεκτική θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τέτοιες περιπτώσεις διαφορών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντελβό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Φαντάζομαι ότι οι συστάσεις σας είναι κάποιες βραχυπρόθεσμες και κάποιες άλλες ε, μακροπρόθεσμες. Σε ό,τι αφορά το Διεθνές Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δικαστήριο. Είπατε ότι θα μπορούσε να ανταγωνιστεί άλλα διεθνή δικαστήρια. Αναφερθήκατε στην Κίνα, στη Σιγκαπούρη. Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες ε, για το πώς θα λειτουργήσει, πώς λειτουργεί μάλλον κάτι τέτοιο σε άλλες υπήρους. Και η δεύτερη μου παρατήρηση αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα. Γιατί είναι ίσονο σημασία και σε αυτό το σημείο, οπότε θα μπορούσατε να βελτιωθεί η πρόσβαση στα δεδομένα. έχετε κάποια άποψη για την ε, δικαιοσύνη πρόβλεψης, δηλαδή όταν έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη και έχουμε μια κοινή βάση δεδομένων, όπου εκεί αποθηκεύονται όλες οι αποφάσεις, ε, υπάρχει κίνδυνος, γι' αυτό ή μας βοηθάει να έχουμε μεγαλύτερη προβλεψιμότητα. Έχετε άποψη για το θέμα αυτό. Γιατί διαβάζω πολλά υπέρ και κατά και προσπαθώ να αποφασίσω για το θέμα αυτό. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Παρακαλώ να σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε. Μικρόφωνο παρακαλούμε για την ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσες ε, ερωτήσεις που θέτουν και προκλήσεις και θα προσπαθήσω να τις απαντήσω στον περιορισμένο χρόνο που έχω. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τις ερωτήσεις του κυρίου Λεμπρετών Το πρώτο σας σχόλιο, αν σας κατάλαβα καλά, αφορά την σύσταση ειδικών δικαστηρίων και τμήματων στα κρατη Αν σας κατάλαβα καλά, είπατε ότι είχατε αμφιβολίες για το αν η σύσταση δικαστηρίων είναι καλή ιδέα, αλλά είπατε ότι η σύσταση ειδικών τμήματων θα ήταν ε, ένας εφικτός δρόμος προς τα μπρος. Εδώ θα το άφηνα εντελώς αυτό στα κράτη-μέλη, το πώς θα εφαρμόσουν την απέτηση να παρέχουν ειδικά δικαστήρια ε, για τους διαδίκους σε εμπορικέ διαφορές. Θα μπορούσαμε να έχουμε είτε ένα ειδικό δικαστήριο είτε ένα ειδικό τμήμα, αναλόγως με το τι ταιριάζει καλύτερα στο δικαστικό σύστημα του κράτους μέλους μπορούσα να φανταστώ, παραδείγματο χάρη κάτω χώρε ε, που εργάζονται τώρα για τη ε, δημιουργία ενό διεθνού δικαστηρίου, θα ήθελαν αυτό το δικαστήριο να το διορίσουν ε, ως το αρμόδιο δικαστήριο για διεθνείς διαφορές. Ενώ η Γερμανία και η Γαλλία που πρόσφατα έχουν συστήσει ειδικά τμήματα, θα ήθελαν να ορίσουν αυτά τα τμήματα. Θα το άφηνα λοιπόν στα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι αυτά τα νέα τμήματα, δικαστήρια, ταιριάζουν στις υφιστάμενες δικαστικές δομές. Σε ό,τι αφορά τώρα τη γλώσσα της διαδικασίας. Βεβαίως αυτή είναι μια τεράστια συζήτηση. Δηλαδή, πώς θα απαντήσουμε το δύσκολο ερώτημα αν πρέπει να επιτρέψουμε διαδικασία στα αγγλικά και κράτη-μέλη που έχουν εισαγάγει διαδικασία στα αγγλικά πρόσφατα είχαν πολύ μεγάλες συνταγματικές συζητήσεις για το θέμα αυτό. Όσο παρακολούθησα εγώ τη συζήτηση και την παρακολούθησα στη Γερμανία, στη Γαλλία και στις χώρες, θεωρώ ότι συνταγματικά δεν αποτελεί πρόβλημα να επιτρέψεις διαδικασίες στην αγγλική γλώσσα για τέτοιες ειδικέ διασυνοριακές υποθέσεις, στο βαθμό που διασφαλίζεται ότι υπάρχει διερμηνία στην πρωτότυπη γλώσσα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι λειτουργούν τα δικαστήρια αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Έχουμε ένα νέο τμήμα στο εφετείο στο Παρίσι που παρέχει διερμηνία στα γαλλικά, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι τα συνταγματικά δικαιώματα όλων των διαδίκων αλλά και του κοινού διασφαλίζονται. Ναι, νομίζω ότι ορθά το, το θέμα είναι πρόβλημα, αλλά αν δείτε τι συμβαίνει στα κρατη θα δείτε ότι υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί αυτό το σημαντικό θέμα. Το ερώτησή σα ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δικαστήριο. Αυτό το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δικαστήριο σε καμία περίπτωση δεν θα αντικαταστήσει τα δικαστήρια των κρατών μελών. Θα συμπληρώσει τα δικαστήρια των κρατών μελών. Συχνά ε, θα αποτελεί ένα πρόσθετο δικαστήριο για τα μέρη σε ό,τι αφορά την δικαιοδοσία μεταξύ του Ευρωπαϊκού, Δικαστικού, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και των Δικαστηρίων των Κρατών Μελών, αυτό θα φεθεί στους διαδίκους. Οι διάδικοι θα αποφασίσουν πού θέλουν, σε ποιο δικαστήριο θέλουν να προσφύγουν. Μπορεί να επιλέξουν το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δικαστήριο, αλλά μπορεί και να επιλέξουν να στραφούν σε ένα δικαστήριο στο κάποιο κράτος μέλος. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν θα έχει υποχρεωτική δικαιοδοσία. Έτσι λοιπόν οι διάδικοι δεν θα παραπέμπονται υποχρεωτικά στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δικαστήριο, αλλά αυτό το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δικαστήριο ε, θα αφήνει τη δυνατότητα στους διαδίκους να αποφασίσουν ποιο είναι ε, το καλύτερο δικαστήριο για να επιλύσουν τις διαφορές τους και πολλά μέρη πιστεύω ότι θα προτιμούν να επιλύσουν τις διαφορές τους στα κράτη-μέλη, στα ειδικά δικαστήρια ενώ άλλα μέρη μπορεί να τίνουν να αναζητήσουν τη δικαιοσύνη σε ένα διεθνές δικαστήριο. Αλλά εγώ θα το αφήνω να το αποφασίσουν οι διάδικοι αυτό. Είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δικαστήριο να συμπληρώνει και όχι να αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τα δικαστήρια των κρατών μελών. Η τελευταία σας παρτήρηση αφορούσε την επιλογή του δικαίου. Στη μελέτη μου περιέγραψα ότι ο, κανο, ο κανονισμός Ρώμη 1 έχει μια ελευθερία στάση σε ό,τι αφορά την ε, επιλογή του δικαίου. μπορεί μπορεί μέρη μπορούν να επιλέξουν ενώ υπάρχουν δύο περιορισμοί στη Ρώμη 1 και εγώ συνιστώ στη μελέτη μου να αρθούν οι περιορισμοί αυτοί για διάφορους λόγους. Κυρίως ε, γιατί δεν ε, προωθούν την επιλογή ενός δικαστηρίου σε ένα κράτος μέλος, αλλά σπρώχνουν τους διαδίκους μακριά από τα κράτη-μέλη και νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν εξυπηρετεί το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, εγώ συνιστώ να έρθουν οι περιορισμοί αυτοί έτσι ώστε οι εμπορικοί διάδικοι να μπορούν ελεύθερα να ασκήσουν την επιλογή τους. Και προχωρώ τώρα στην κυρία Κάφμαν και τις ερωτήσεις της σε σχετικά με τη διαπραγματευτική ισχύ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και έχετε δίκιο. Στην αρχή της μελέτης μου είπα ότι ε, βασίζομαστε στην υπόθεση ότι μιλάμε για εμπορικά μέρη με ίση ισχύ. Τώρα, σωστά είπατε ότι ακόμη και αν δούμε τις εμπορικές σχέσεις, Πολύ συχνά έχουμε σχέση όπου ένας έχει, είναι σε ισχυρότερη θέση, ε, οι μικρές ε, εταιρείε ε, έναντι ε, μεγάλων εταιριών ή για άλλους λόγους. Φυσικά στις εμπορικές σχέσεις βλέπουμε ότι οι διάδικοι δεν έχουν την ίδια την πραγματική ισχύ. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζεις αυτές τις καταστάσεις από κανονιστική σκοπιά. Και εδώ γίνεται προβληματικό. Γιατί δεν μιλάμε για τις εμπορικές σχέσεις είναι σχετικά δύσκολο εκ των πρότερων να πεις ποιο μέρος θα είναι το ισχυρότερο. Μπορεί να είναι το μεγαλύτερο μέρος, αλλά μπορεί να είναι και το μικρότερο που θέτει τους όρους. Και μπορεί να είναι το μέρος που έχει το μεγάλο μερίδιο στην αγορά, αλλά μπορεί να είναι και το αντίστροφο. Έτσι λοιπόν από κανονιστική σκοπιά είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις ε, αυτή την κατάσταση. Όταν μιλάμε για καταναλωτικές συμβάσεις, εκεί είναι διαφορετική κατάσταση, γιατί μπορούμε να υποθέσουμε ότι σε πιο δύναμη θέση είναι ο καταναλωτής. Αλλά δηλαδή, όταν μιλάμε για εμπορικές συμβάσεις είναι πιο δύσκολο. Επομένως, πώς θα διασφάλιζα ότι τα δικαιώματα των πιο αδύναμων μερών, εμπορικών μερών, των μικρών εταιριών, παραδείγματο χάρη, προφυλάσσονται. Εγώ θα συνιστούσα το εξή. Θα διασφάλισα ότι σε όλε τι προτάσει που καταθέτω θα πρέπει να διασφαλίσουμε όλα τα συνταγματικά δικαιώματα, δηλαδή να προσφέρουμε στα μέρη το δικαίωμα κράση στο δικαστήριο, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Νομίζω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σε μία επιταχυμένη διαδικασία γίνονται σεβαστά όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα, όλες οι συνταγματικές απαιτήσει. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα των μερών, τα θεμελιώδη δικαιώματα, δεν θυσιάζονται στο βωμό τη ταχύτητα και τη αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι μικρότερε εταιρείε ή εταιρείε για άλλου λόγους βρίσκονται σε πιο αδύναμη θέση, προστατεύονται καλά. Στο ευρωπαϊκό μελλοντικό Καθεστώ. Ελπίζω να σα απάντησα. Τώρα, στις ε, δικές σας ερωτήσεις για το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δικαστήριο και τις σχέσεις με τα άλλα διεθνή δικαστήρια. Τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε δει παγκοσμίω ότι χώρε προσπαθούν ε, να συστήσουν διεθνή εμπορικά δικαστήρια προκειμένου να προσελκύσουν τι διεθνεί εμπορικέ διαφορέ. Ένα μεγάλο όγκο εμπορικών διαφορών. Και όλα αυτά τα διεθνή δικαστήρια προσπαθούν να είναι τόσο ελκυστικά όσο εκλογιστικά γίνεται για τα διεθνή μέρη, για τους διεθνείς διαδίκους και προσπαθούν να προσελκύσουν διαδίκους από διάφορες δικαιοδοσίες και από διάσημες δικαιοδοσίες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν δείτε το δικαστήριο στο Ντουμπάι, παραδείγματος χάρη, βασικά ε, εκεί εργάζονται πρώην δικαστές από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, έτσι λοιπόν νομίζω ότι ήρθε ο καιρό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι. Γιατί δεν έχω αμφιβολία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθ' ω κοινότητα των κρατών μελών έχει τα ίδια να προσφέρει στου διεθνεί διαδίκους, αν όχι περισσότερα, λόγω τη επικλομορφίας ε, που έρχεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με τα υπόλοιπα διεθνή εμπορικά δικαστήρια. Το δεύτερο σχολείο σα αναφέρθηκε στην πρόσβαση στα δεδομένα. Το αναφέρω και εγώ στη μελέτη μου ότι οι δικαστές όταν ε, έχουν να κάνουν διασυνοριακές υποθέσεις στην πράξη, οι εθνικοί δικαστές έχουν δυσκολία πρόσβασης ε, στα δεδομένα, κυρίως ε, όταν τα δεδομένα αυτά σχετίζονται με το ελλαδοπό δίκαιο ή έχουν δυσκολίες πρόσβαση σε υποθέσεις που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η πρότασή μου βασικά συνιστάται στο να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Τώρα για το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει, δεν το ξέρω, δεν το ερεύνησα αυτό. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να διερευνηθεί για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για να βελτιώσουμε το έργο των δικαστών και το αποτέλεσμα των ε, διαδικασιών να είναι πιο προβλέψιμο. Δεν το κάλυψε αυτό στη μελέτη μου γιατί ήταν εκτός του πεδίου εφαρμογή, αλλά νομίζω ότι θα άξιζε να διερευνήσουμε την ε, δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης λεπτομερέστερα, ίσως στο πλαίσιο μιας άλλης μελέτης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και για τις απαντήσεις σας. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο και να καλωσορίσω ταυτόχρονα την Δ. Τατιάνα Εύας από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Ερευνών, η οποία θα μας παρουσιάσει την ε, αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας στην ταχεία επίλυση εμπορικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Εύας, έχετε 15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρούλ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Νομίζω θέσατε τις βάσεις για τη ε, συνέχεια της συζήτησης και αναφερθήκατε στις ε, επιπτώσεις. Εγώ θα εστιάσω στα οικονομικά ωφέλη και είναι ε, λογική η ακολουθία της σκέψης αυτής. Συνεχίζοντας λοιπόν από την προηγούμενη παρουσίαση, θα χρησιμοποιήσω την ε, προσέγγιση της αγοράς για να παρουσιάσω ποια είναι τα οικονομικά ωφέλη μέσω της ευρωπαϊκής συγκέντρωση επίλυση διαφορών. Ποια είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία λοιπόν στην επίλυση εμπορικών διαφορών. Η παρουσίασή μου χωρίζεται σε πέντε κύρια σημεία, πέντε βήματα. Ξεκινάμε με μια ερώτηση. Γιατί λοιπόν χρειάζεται να αναλάβουμε δράση από εμπορική σκοπιά. Τι σημαίνει αυτό για την αγορά. Θα σας εξηγήσω πρώτα τι διακυβεύεται, σε τι πόσο ανέρχεται η αξία της ε, διαδικασίας επίλυσης διαφορών, τι βήματα μπορούν να γίνουν για να βελτιωθούν οι επιδόσεις στην αγορά αυτή. Και τέλος, θα εστιάσω στα ωφέλη που μπορούμε να έχουμε εάν αναλάβουμε δράση σε αυτόν τον τομέα. Και συμπερασματικά θα επιστρέψω στο γιατί και ελπίζω μέχρι τότε να είναι σαφής η απάντηση. Θα ξεκινήσω λοιπόν και θα αναφερθώ στην αγορά. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τις διαφάνειες. Ξεκινάμε λοιπόν με το γιατί γιατί λοιπόν είναι σημαντικό να εξετάσουμε το ερώτημα αυτό από την ε, οπτική του εμπορίου, της αγοράς. Ας δούμε τη δομή της αγοράς. Χαρακτηρίζεται από ανταγωνιστικότητα, από σαφήνεια και από το κόστος. Ανταγωνιστικότητα. Όπως αναφέρθηκε, η Ευρώπη βρίσκεται σε ανταγωνισμό με τις άλλες περιοχές του κόσμου και κοιτάζοντας την δομή των αγορών βλέπουμε ότι η αγορά επίλυσης διαφορών χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση, ψηφιοποίηση και ανταγωνισμό ανάμεσα στα ε, κράτη. Υπάρχουν ορισμένοι πολύ σημαντικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τη δομή της αγοράς και χρειάζεται λοιπόν να δείξουμε προσοχή. Το κυριότερο επιχείρημα είναι ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναλάβει συλλογική δράση, οι ευκαιρίες που δημιουργεί αυτή η αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα θα χαθούν. Έπειτα, γιατί γιατί να αναλάβουμε δράση. Αυξάνοντας την σαφήνεια θα μειώσουμε το κόστος, το κόστος της επίλυσης διαφορών που με τη σειρά του θα καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ελκυστική για την επίλυση εμπορικών διαφορών. Υπάρχει αρκετά καλή εμπειρία με την εναρμόνιση των κανόνων ουσιαστικού δικαίου αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη βιομηχανία είναι πάρα πολύ θετική. Χαρακτηρίστηκε μάλιστα η πρωτοβουλία αυτή ως μία από τις σημαντικότερες των τελευταίων 30 ετών. Όμω, μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα από την οικονομική άποψη και αυτό θα αποφέρει ωφέλη στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μετά, θα ασχοληθούμε και με το κόστος στην παρουσίαση οι καθυστερήσεις εκδίκας αποφάσεων ε, επιφέρουν πρόσθετο κόστος, γι' αυτό λοιπόν η ταχεία διαδικασία θα έχει οικονομικά ωφέλη. Περνάμε στο επόμενο σημείο, η αγορά και το μέγεθος αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά ανταγωνιστική. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη των 28 είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο σε ό,τι αφορά τις νομικές υπηρεσίες και η αγορά επίλυσης διαφορών ανέρχεται στα 226 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Βλέπετε πως τα ποσά είναι τεράστια λοιπόν, η αγορά είναι μεγάλη, οπότε σίγουρα μπορούμε να διερευνήσουμε περισσότερο την κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει το 22% της παγκόσμιας αγοράς. Τώρα, ε, σε ό,τι φορά την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα, η η αξία της ε, αγοράς επίλυσης διαφορών έρχεται στα 51 δισεκατομμύρια ευρώ και η εμπορική επίλυση διαφορών business to business ανέρχεται περίπου στα 24,5 δισεκατομμύρια και οι διασυνοριακές υποθέσεις 8,1. Η καθηγήτρια κυρία Ρούλε μας είπε ήδη πως είναι άνηση η κατανομή του ποσού αυτού ε, εδώ βλέπετε το ποσοστό του ΑΕΠ της κάθε χώρας και το μερίδιο που έχει η κάθε χώρα στην αγορά νομικών υπηρεσιών. Γιατί όμως αναφέρω αυτά τα στοιχεία και τα συσχετίζω στην ε, μελέτη μου. Στη βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα αυτό, το ΑΕΠ μπορεί να ε, είναι ενδεικτικό του μεριδίου της αγοράς. Βλέπουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία είναι στις πρώτες θέσεις. Τώρα τι διακυβεύεται. Πολλά. Η αγορά επίλυσης ε, διαφορών μπορεί να αποφέρει σημαντικά έσοδα, όμως αυτή τη στιγμή, όπως ακούσαμε, δεν υπάρχει ίση κατανομή στα κράτη-μέλη. Εδώ περνάμε στο επόμενο ερώτημα και στην επόμενη διαφάνεια. Τι μπορούμε δηλαδή να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα όχι μόνο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εντός όπως ανέφερα ήδη, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την απόφαση εκδίκασης μιας ε, διαφοράς και της επιλογής δικαιοδοσίας. Οι τρεις κυριότεροι παράγοντες που αναφέρονται στην ε, πιο πρόσφατη έρευνα από το 2007 της Boston Consulting Group είναι οι εξής. ο περίπλοκος χαρακτήρας και οι μακροχρόνιες διαδικασίες, η εμπειρία των δικαστών και η ταχύτητα της ε, διαδικασίας. Για το τελευταίο, ο χρόνος εκδίκασης είναι ένας από τους πέντε κυριότερους ε, λόγους επιλογής. Γι' αυτό τα ωφέλη στην αγορά εστιάζουν περισσότερο στην ταχύτητα της διαδικασίας. Είναι ένα από τα κυριότερα στοιχεία. Σίγουρα δεν είναι το μόνο στοιχείο, η μόνη λύση, όμως ε, είναι πολύ σημαντικό, είναι κέρια σημασίας για την ε, επιλογή, για τη δομή της αγοράς. Το γιατί δηλαδή οι διάδικοι αποφασίζουν να εκδικάσουν μια απόφαση σε συγκεκριμένες δικαιοδοσίες. Τώρα, ο χρόνος, γιατί είναι τόσο σημαντικός. Διότι Φαίνεται από την ε, σχετική βιβλιογραφία ότι οι μακροχρόνιες δίκες υπονομεύουν την ε, ασφάλεια, τη βεβαιότητα των συναλλαγών και ε, συνοδεύονται από υψηλό κόστος. Σε αυτό θα μπούμε σε λεπτομέρειες στη συνέχεια. Τι μπορεί τώρα να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί μέσω συλλογικής δράσης να μειώσει τις καθυστερήσεις για να απολαμβάνουμε τα ωφέλη της ταχείας διαδικασίας απειλής διαφορών. Και ως απόρρια αυτού τι μπορούμε να κάνουμε λαμβάνοντας δράση. Ποια είναι τα ωφέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια είναι η προστιθέμενη αξία. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, αναπτύξαμε ένα μοντέλο μέσα στη μελέτη, το οποίο έχει δύο ε, πτυχές. Πρώτον, κοιτάζει την ε, μείωση του κόστους, δηλαδή με απλά λόγια πόσο μπορούμε να εξοικονομήσουμε εάν ε, μειωθεί ο χρόνος εκδίκασης. Και δεύτερον, πόση δουλειά μπορούμε να προσελκύσουμε, πόσες υποθέσεις επίλυσης διαφορών μπορούμε να προσελκύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εάν το σύστημα ε, γίνει ταχύτερο. Για να κάνουμε αυτούς τους υπολογισμούς, συνδυάσαμε τον άμεσο αντίκτυπο ε, του κόστους, μετά το γενικότερο αντίκτυπο στην Ευρωπαϊ... στην οικονομία της Ένωσης και τη συνολική οικονομική αξία. Αυτά τα τρία στοιχεία θα σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε τα νούμερα που θα δείτε στη συνέχεια. Μετά βλέπετε την γενικότερη δομή. Ας κοιτάξουμε το πρώτο στοιχείο. Πόσα χρήματα δηλαδή μπορεί κάποιος να κερδίσει εάν μειώσει την ε, διαδικασία, το χρόνο της ε, διαδικασίας εκδίκασης. Έχουμε τρεις περιπτώσεις στη μελέτη που εξετάζουν ε, τρεις περιπτώσεις μείωσης του χρόνου. Τρεις μεγάλοι παράγοντες ποσοτικοποίησης, το ποσό που διακυβεύεται, η μείωση του χρόνου και τα διαφυγόντα κέρδη. Πρώτον, στην πρώτη περίπτωση υπολογίζεται ότι είναι περίπου 30 δισεκατομμύρια το χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 ε, το κόστος ε, της εκδίκασης μιας υπόθεσης. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνει το κόστος, την αμοιβή των ε, δικηγόρων, αλλά μόνο τα έξοδα, τα δικαστικά έξοδα. Τώρα, τα, τώρα οι διάδικοι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό το ποσό, διότι αυτό το ποσό ε, είναι προς εκδίκαση. Πολλές φορές η δέσμευση διαρκεί πάνω από... Ε, το πάγωμα διαρκεί πάνω από μέχρι 150 ημέρες στην περίπτωση της Λιθουανίας, όμως σε κάποιες χώρες όπως η Ελλάδα το πάγωμα μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 5 χρόνια. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δούμε τρεις ε, περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση προσπαθούμε να φέρουμε όλα τα κράτη-μέλη στο μέσο όρο, δηλαδή στις 196 μέρες παγωματός. Το δεύτερο σενάριο, όλα τα κράτη-μέλη να έχουν σε πρώτο στάδιο ε, ανώτατο όριο 6 μηνών και το τρίτο σενάριο αν όλες οι διαφορές επιλύονται στο χρονικό διάστημα των 25 καλύτερων με αυτήν την έννοια δικαιοδοσιών. Η πρώτη περίπτωση που είναι λιγότερο φιλόδοξη θα έχει κέρδος 2,1 δισεκατομμυρίων το χρόνο, η δεύτερη περίπτωση 2,4 και η τρίτη 3 δισεκατομμύρια ετησίως. Αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Η επίσπευση της διαδικασίας δεν είναι κάτι το αδύνατον, ούτε συνεπάγεται θέσπιση νέων ε, δομών και κανόνων. Θα μπούμε όμως ε, στη συνέχεια σε λεπτομέρειε ό,τι αφορά τις παραμέτρους που χρησιμοποίησαμε για να υπολογίσουμε και να φτάσουμε σε αυτά τα στοιχεία. Έπειτα, η αξιολόγησή μας εξετάζει το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσέλκυση ε, νέων υποθέσεων. Εδώ πάλι υπάρχουν τρεις υποθέσεις που εξετάσαμε. Η μία είναι πιο συντηρητική, χρησιμοποιεί τις υφιστάμενες δομές, είναι μικρή η αύξηση και η τρίτη περίπτωση που εξετάσαμε είναι η πιο φιλόδοξη που απαιτεί μεγάλες αλλαγές στην ε, αγορά ε, εκδικαστή φορών. Κοιτάξαμε τη σχέση ανάμεσα στο ΑΕΠ και της ε, παροχή νομικών και την παροχή νομικών υπηρεσιών και στην περίπτωση business to business και προσπαθήσαμε να υπολογίσουμε τα στοιχεία για την κάθε περίπτωση. Το πιο μετριοπαθές ας πούμε σενάριο θα ε, δημιουργήσει κέρδη 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και το πιο φιλόδοξο 2,7 Συμπερασματικά. Επανέρχομαι στο αρχικό μου ερώτημα. Τι μπορεί δηλαδή να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι έχει να κερδίσει. Βασισμένη λοιπόν σε αυτά τα στοιχεία τα οποία μπόρεσα μόνο πολύ συνοπτικά να σας εξηγήσω, εάν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει βήματα προς ε, επίσπευση της διαδικασίας, θα μπορέσουμε πλέον να κάνουμε λόγο για κέρδη 3,7 έως 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Αυτό βέβαια δεν είναι χωρίς ε, μειονεκτήματα, δεν θα γίνει αμέσως και απαιτεί την λήψη αρκετών μέτρων, δέσμης μέτρων, όμως ε, είναι εφικτό. Επίσης, το νούμερο αυτό που σας ανέφερα είναι, μία, είναι, είναι αρκετά ε, μετριοπαθές. Προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε στα κατώτατα όρια και δεν συμπεριλάβαμε διάφορες ε, περιπτώσεις, για παράδειγμα, της δικαστικής συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη ή διαδικασίες ε, κατάρτισης. Όμως, ήταν πραγματική αποκάλυψη αυτά τα στοιχεία και νομίζω πως η απάντηση ε, στο γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ε, επισπεύσει τις διαδικασίες επίλυσης εφορών είναι προφανής. Η μέθοδος που χρησιμοποίησαμε βρίσκεται στο τέλος της μελέτης, γι' αυτό λοιπόν ε, σας παρατρύνω να την διαβάσετε, να κοιτάξετε και τους συνδέσμους και φυσικά είμαι ανοιχτή σε ερωτήσεις και σχόλια και με χαρά μου θα συμμετέχω στην συζήτηση που θα ακολουθήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Υπάρχουν ερωτήσεις από τους βουλευτές. Κυρία Νίμπλερ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Δύο ερωτήσει έχω μόνο για, για να διευκρινιστούν κάποια πράγματα. Πρώτον, μας είπατε ότι ε, η διάρκεια, χρονική διάρκεια επίλυση σε μια διαδικασία έχει να κάνει και με το πόσο ελκυστική είναι. Αυτό βέβαια μου φαίνεται κάπως... Ε, απλή, κάπως απλώς αναπάντηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες και είναι πολύ πιο πολύ περίπλοκο το ζήτημα. Ε, έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες των ε, διαδίκων. Δεν μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τόσο εύκολα ε, την κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν εσείς που βασιστήκατε για να μας παρουσιάσετε αυτά τα στοιχεία. Έπειτα, σε ό,τι αφορά το Brexit, η 31η Μαΐου πλησιάζει. Έχετε λοιπόν κάποια εικόνα του πώς μπορεί να διαμορφωθεί το σκηνικό και ο ρόλος του Ηνωμένου Βασιλείου στην αγορά αυτή. Σας ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε σε ερωτήσεις παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Ε, προσπαθώντας ε, να εξετάσουμε τα δεδομένα που έχουμε, ε, ενοποιούμε δεδομένα και για τις πιο σύντομες ε, δίκες, αλλά μόνο αστικές και εμπορικές. Μέσο όρο για τα 20 και κράτη είναι 273 ημέρες ο μέσος όρος διάρκειας μιας δίκης. Αστικής και εμπορικής, 50% λοιπόν των τρεχών δικαιοδοσιών, αν πάρουμε με την υπόθεση ότι και πιο περίπλοκες αλλά και πιο απλές ε, δίκες έχουν να κρίνουν, τότε θα πρέπει να μπορεί και το υπόλοιπο 50%. Όπως είπα, πρόκειται για υπολογισμό ε, ενοποιημένο, αλλά μας δίνει μια ένδειξη. Προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε δύο διαφορετικούς δείκτες από επιχειρήσεις στην Ευρώπη και από μια μελέτη του Συμβουλίου της Ευρώπης που παρακολουθεί τη διάρκεια εκδίκασης μιας υπόθεσης από το δικαστήριο. Οπότε θα ήταν και πιο υψηλή η αριθμή, η διάρκεια δηλαδή. Ε, και όπως είπα έχουμε πολύ συντηρητικά στοιχεία κοιτώντας μόνο την πρωτόδικη απόφαση. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα ήταν μειωτική η τάση. «296 μέρες ψεύω εγώ θα ήταν ε, αυτή τη στιγμή μια λογική υπόθεση για ένα μέσο όρο, λαμβανόμενο υπόψη και το πιο περίπλοκο ε, δικών. Επίσης μιλάτε για την ποσοστοποίηση μας και το μερίδιο αγοράς που έχω δείξει και την αύξηση 10, 12, 20%. Αυτό στηρίζεται στην υπόθεση της αποχώρησης από, την Ευρωπαϊκή Ένωση του Βασιλείου. Ελαστικότητα της αγοράς και σύνολο με την υπόθεση ότι θα μπορέσει να προσελκύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να αυξήσει έτσι το μεριδιό της σε δίκες μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει στήσει άλλο συνάδελφος ε, το λόγο για να υποβάλει ερωτήσει. Σας ευχαριστώ λοιπόν και τις δύο μιλητριές μας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσε πληροφορίε. Ευχαριστώ πολύ. Και συνεχίζω με το σημείο 18 στην ημερήσια διάταξη. έχουμε να κάνουμε με την συλλογική αποκατάσταση δικαιωμάτων. Ε, πρώτα έχουμε μια παρουσίαση μελέτης και μετά θα ακούσουμε ειδικού με συζήτηση υπό τη μορφή ακροάσεως. Στο πλαίσιο της δουλειάς μας της κοινοβουλευτικής σε μια πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για οδηγία σχετική με την ε, αποζημίωση για ηθική βλάβη ή άλλες κυρωτικές αποζημιώσεις προς, το, προς των καταναλωτών. Ένα New Deal για τους καταναλωτές. Ήταν αυτό το οποίο είχε προβλέψει με το πρόγραμμα εργασίας της το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της προσαγωγής και ε, περιορισμό των συνεπειών της παράβασης του ευρωπαϊκού δικαίου με την αποκατάσταση των ε, καταναλωτών στα δικαιώματά τους. Έτσι λοιπόν ξεκινούμε με την παρουσίαση της μελέτης. Η Επιτροπή μας δηλαδή είχε ζητήσει από το Policy Department για τα δικαιώματα των πολιτών και τις θεματικές υποθέσεις μία μελέτη για την ε, συλλογική αποκατάσταση στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο εκ των συντακτών είναι σήμερα εδώ και θα μας παρουσιάσουν την ε, μελέτη τους. Η καθηγήτρια Φαμπιέν Ζολτσεσέκ, πρώτα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Versailles Saint-Quentin της Γαλλίας. Και η κυρία, η καθηγήτρια Μαρία Χωσέα Σαμπότ, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Παρίσιου του, παρά τη Γαλλία. Θα σας παρακαλώσω λοιπόν να λάβετε το λόγο, κυρίες μου, συνολικά για 15 λεπτά, για να έχουμε μετά και το χρόνο για τις ερωτήσεις του συναδέλφων, Ποιος θέλει να ξεκινήσει, ποια θέλει να ξεκινήσει. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ που μα δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τη μελέτη τη Ένωση των Σοχοπεξπέρ των τελευταίων μηνών. Η παρουσίαση θα γίνει και ολοκληρή στα γαλλικά. Η συνάδελφος Μαρία Ζωζέ Ραζάρμπο θα κάνει το πρώτο, πρώτο μέρος της παρουσίαση. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, Μεγάλη τιμή για μένα η ευκαιρία να σας παρουσιάσω σήμερα εδώ την μελέτη μας στο πλαίσιο του δικτύου Τρόνσο Ξέχ μαζί με τον Ραφαέλ Αμαρό, την Φρεντερίκ Βαρκοσόν και άλλους που έχει να κάνει με την συλλογική αποκατάσταση δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στηριζόμαστε πρώτα απ' όλα σε κανονισμούς, οδηγίες, συστάσεις, ε, ψηφίσματα, αποφάσεις, δηλαδή νομοθετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνωρίζουν την ανάγκη να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα της συλλογικής αποκατασταση, για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η καλύτερη απόδοση αυτής. Πρέπει επίση να σημειώσουμε ότι οι συλλογικέ αγωγέ ε, βελτιώνουν την ασφάλεια δικτύου για, ε, για όλα τα υποκείμενα δικαίου και όχι μόνο για τα θύματα ή για τους ε, ζημιοθέντες. Μπορεί δηλαδή να προστατεύσει τις επιχειρήσεις και κατά του κινδύνου ενός forum shopping που έχει μετατρέψει, όπως άλλωστε αποδεικνύει και η υπόθεση Βέντη της ΗΠΑ, σε ένα πόλο έλξης για τη διευθέτηση δικαστικών διαφορών. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πτυχές που μπορούν να προβληθούν περισσότερο, ώστε να ε, καταστεί ακόμη πιο ελκυστικό αυτό το όμορφο εγχείρημα που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ε, εγκυρότητα της μελέτης μας. Καταρχάς έχει καταρτιστεί με βάση τις ε, τοποθετήσεις της 25ης Ιανουαρίου του 2018 στη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή, Ένωση, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενόψη της σύστασης για ένα κοινό καθεστώς για τις συλλογικές αγωγές αποκατάστασης και αποζημίωσης, απουσία μέσων προστασίας που μπορεί να έχουν δυσμενή αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην ιστορική αγορά και άρα να εμποδίσουν έτσι την ανάπτυξη αυτή σε όρους οικονομικούς και κοινωνικούς. Επίσης ε, παρακολουθούμε και την ε, θεωρία του συγκριτικού δικαίου που μας ενδιαφέρει ως ε, ερευνήτρες και βέβαια είναι ιδιαίτερος λόγω και του γεγονός ότι ήμουν δικηγόρος με ιδιαίτερη ανασχόληση στα θέματα των συλλογικών αγωγών και επίσης έχουμε και δύο κείμενα στο παράρτημα που καταγράφουν πολύ ενδιαφέρουσε εμπειρίες σε σχέση με την άνεση εξέλιξη παιδοκράτων μελών για τις συλλογικές αγωγές αποζημίωσης. Κάποια κρατημέλη έχουν υιοθετήσει τη σχετική, στη δική του ενωμή τάξη τα σχετικά νομοθετήματα, πράγμα το οποίο ήταν ε, απίθανο μερικά χρόνια ακόμη πριν. Ορισμένα όμω ακόμη δεν έχουν προχωρήσει και αναμένεται τη δράση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω εκ τούτου έρχεται εν ευθέτω χρόνο, γιατί φαίνεται ότι τα κρατη είναι διτεθειμένα να παρακολουθήσουν την, το εξελισσόμενο ρεύμα το αναδεικνύωμενο ρεύμα, γιατί θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη που του επιτρέπει να ξεπεράσουν τα πολιτικά εμπόδια με τα οποία είναι αντιμέτωπα. Και έτσι. Με τη βάση αυτή που σας ανέφερα, εξετάσαμε την ε, πρόταση οδηγίας για την συλλογική αγωγή και που σας παρουσιάζουμε καταρχάς με βάση τις ε, διατάξεις που θεωρούμε ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν λόγω και των αποκλήσεων ως προς τα δικονομικά ζητήματα μεταξύ κρατών μελών. Δεύτερον, τους κανόνες που, έχουν, ε, που απαιτούν κάποιες διευθετήσεις, κάποιες ρυθμίσεις και τρίτον τους κανόνες εκείνους της διατάξεις που ακόμη δεν έχουν καλυφθεί γιατί δεν έχουν προβληθεί από την πρόταση. Προτάσεις λοιπόν θα πρέ... που θα πρέπει ιδιαίτερα να εξετάσουν την υιοθέτηση ενός μηχανισμού συλλογικής ε, αγωγής που να εξασφαλίσουν τις δύο αποκαταστάσεις, δηλαδή την πάυση της ε, ζημιογόνου ε, συμπεριφοράς ή κατάστασης και την αποκατάσταση της ζημίας. Έχουμε να κάνουμε με αποζημίωση, με μια πρόταση που θα πρέπει να υποστηριχθεί, για να, γιατί δεν θα ήταν καλό να, ενταχθούν, να εισαχθούν στις εθνικές αερομες τάξεις περιορισμοί σε αυτήν που ενδεχομένω θα οδηγούσαν σε συνολική απαγόρευση των αποζημιώσεων για ηθική βλάβη ή άλλων κυρωτικών αποζημιώσεων. Επίσης, η εκπροσωπευτική αγωγή, όπως ονομάζεται, μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο όρο για την ανάληψη δράση εξ ονόματος μιας ομάδας, αλλά θα μπορούσε να οδηγήσει και σε σύγχυση. Πρόκειται για μια έκφραση που ορισμένα κράτη, όπως διαπιστώνουμε, έχουν ακολουθήσει και κατά την ε, επεξεργασία ε, αγωγών για πάυση ενέργειας ή ε, παράληψης. Ενώ η συλλογική αγωγή είναι ένας ευρωπαϊκός όρος και μπορεί να καλύψει και την ε, διάσταση της ε, αποζημίωσης, δηλαδή και η πάυση της ε, πράξης υπαράληψης, αλλά και η αποκατάσταση των, ζημιών είναι αυτό που ζητείται από έναν αριθμό συγκεκριμένων ή μη ατόμων και άρα έχουμε να κάνουμε με μια συλλογική αγωγή. Πεδίο φαρμακής. Αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης, καθώς το παράρτημα αναφέρεται σε 59 ευρωπαϊκά νομοθετήματα και έτσι καλύπτει ένα ευρύ πεδίο, αλλά η συλλογική αποκατάσταση αναφέρεται σε καταναλωτή ως ιδιώτη, νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο δράσε ε, με ιδιότητα άλλη από αυτή του καταναλωτή ή όπως περιγράφεται γενικά στο κείμενο αποκλείεται από αυτή την συλλογική αγωγή για αποκατάσταση. Και άρα έχουμε να κάνουμε με το follow-on actions που μπορεί να οδηγήσουν σε αρκετό αριθμό δράσεων, αγωγών για την αποκατάσταση δικαιωμάτων θυμάτων που δεν προβλεπόταν το 2014. Μπορεί ο αποκλεισμό αυτό να οδηγήσει και σε διακριτική, να κριθεί ω διακριτική μεταχείριση. Αν μιλούσαμε μόνο για υποκείμενα δικαίου, θα είχαν αυτέ οι αγωγέ ακόμη ευρύτερο πεδίο και δεν θα ήταν απαραίτητο καν το παράρτημα. Έτσι λοιπόν θα ήταν το νομοθέτημα προσαρμοσμένο στη σύγχρονη εποχή. Θα μετατραπόταν δηλαδή σε ένα εργαλείο κοινωνική δικαιοσύνη. Μεταξύ των ε, κανόνων που πρέπει επίσης να προσέξουμε ιδιαίτερως έχει να κάνει με την ιδιότητα του διαδίκου ή τις προϋποθέσεις για να αναλάβει κανείς την ιδιότητα του διαδίκου, τις προϋποθέσεις για την εγγραφή στον κατάλογο, τις ε, προϋποθέσεις ε, δράσεως μέσα στην αγωγή, ad hoc προϋποθέσεις που βεβαίως μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα και με την ορίμανση στο πεδίο αυτών των κρατών μελών άμεση σχέση μεταξύ των στόχων της οντότητας και των δικαιωμάτων που αποδίδει το σχετικό ευρωπαϊκό δίκαιο, του οποίου η παράβαση θεωρείται ότι οδηγεί στην εν λόγω συλλογική ε, αγωγή, είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός παράγων. Στις διασυνοριακές ε, αγωγές, η αναγνώριση του διαδίκου σε ενώσεις κρατών μελών, από άλλο, ε, κράτου μέλους άλλο από αυτό της δίκης, η δυνατότητα για κοινή δράση και συνεργασία σε μια δίκαιο των διαδίκων της μιας πλευράς των αγώνων δηλαδή έχει πολύ μεγάλη σημασία και αποτελεί σημαντική προόδο. Μπορεί να ενισχυθεί και η έννοια της ε, παρέμβασης και η μετα φορά σε εθνικό κείμενο μπορεί να βελτιώσει ακόμη περισσότερο με διευκρινήσεις ε, το νομοθέτημα. Όταν ε, κάνει μια αναγνωριστική κρίση ο δικαστής, ή, όταν, ε, ή πέραν των περιπτώσεων κατά την οποία είναι υποχρεωτική η αποζημίωση, πρέπει να υποστηρίξουμε αυτές τις ε, προτάσεις. Η δικονομική κανόνας που έχουμε να κάνουμε την ενημέρωση για τις ε, αγωγές του άρθρου 9, το οι συνέπειε των τελικών αποφάσεων άρθρο 10, την άρση της παραγραφής άρθρο 11, της δικονομικής ε, νομιμότητας του, του συστήματος των αποδείξεων, του συστήματος των κυρώσεων και της αρρωγής στους ε, διαδίκους είναι πολύ σημαντικές ε, παράμετροι. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να προσθέσουμε και το άρθρο 3β όπου προβλέπεται ότι η αποζημίωση εναντί ενός κοινού τέτοιου τύπου πάνω απ' όλα υπηρετεί το συμφέρον του καταναλωτή. Άλλοι κανόνες θα ε, απαιτούσαν, θεωρούμε, κάποιες η ε, παραδείγματι, η δικαστική, εξοδικαστική διευθέτηση, η ρύθμιση. Εάν αυτή η πρόνοια διατηρηθεί, θα πρέπει και να ενισχυθεί, αντικαθιστώντας τον προαιρετικό χαρακτήρα από έναν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Και έτσι αντί να λέγεται ότι τα κράτη-μέλη δίνανται να προβλέψουν ή να συνάψουν μια συμφωνία, θα μπορούσαν να υποχρεωθούν τα κράτη να προβλέψουν μηχανισμό που θα επέτρεπε στους διαδίκους να συνάψουν τη συμφωνία και να τους υπαγάγουν σε μια δικαστική υπαγωγή. Στο εδάφιο 4 του άρθρου 4 που δίνεται στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να περιορίσουν σε, ορισμένους, ε, σε ορισμένες ενώσεις προσώπων την χρήση ορισμένων ενδίκων μέσων είναι για μας επικίνδυνος περιορισμός γιατί μπορεί να αποτελέσει και πηγή σημαντικού forum shopping επιλογής, δηλαδή της πιο πρόσφορης δικαιοδοσία. Ευτυχώς το opt-in δεν έχει επιλεγεί ως κανόνας από την πρόταση, αλλά ούτε και ο κανόνας του opt-out. Επομένως οι κανόνες ή, ή μάλλον βασικές αρχές φαίνεται να μην παρακολουθούνται σε όλη τη διάρκεια της προτάσεως. Υπάρχουν κάποιες, ε, υπάρχει ανάγκη να διαβάσουμε και να αναλύσουμε με πολλούς τρόπους και με ερμηνεία ακοντράριο για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Και έτσι υπάρχουν, ε, επί παραδείγματι, υπάρχει πρόβλεψη για υποχρεωτική εντολή ε, ώστε να προβεί κανεί ε, εξ καταναλωτόν των καταναλωτών σε μια αγωγή αποζημίωση. Και αυτό το βλέπουμε και από το άρθρο 6.1 που λέει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να απαιτήσουν εντολή πριν από την έκδοση ετοιμιγορία, όπου η εντολή δεν έχει χρονικό περιορισμό και άρα οι διάδικοι θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε forum shopping, πράγμα επικίνδυνο. Ε, επιλέγουν δηλαδή το κράτος εκείνο στο οποίο η εντολή δεν απαιτείται για την εκκίνηση μιας αγωγής. Επίσης ε, το άρθρο 6.3 που αναφέρεται στην αγωγή ε, που δεν είναι αναγνωριστική για την αποζημίωση με συγκρίσιμη ζημία όπου προβλέπεται ότι δεν μπορεί η εντολή να είναι προϋπόθεση για την κίνηση μιας αγωγής. Αυτό μπορεί επίσης να προβλέπεται μάλλον επίσης και για τις αγωγές χαμηλής αξίας. Η εντολή λοιπόν δεν πρέπει να απαιτείται εδώ γιατί ήταν δυσανάλογο κάτι τέτοιο. Το opt-in που απαιτείται και που προσδιορίζει κάποια όρια, ιδίω για τι χώρε που το έχουν ήδη προβλέψει το σύστημα αυτό. Δεν είναι το προτιμότερο. Εμεί θα προτιμούσαμε ένα μεικτό σύστημα. Ένα σύστημα όπω αυτό του Βελγίου, όπου ο δικαστή μπορεί κατά περίπτωση να επιλέξει την προσφορότερη ρύθμιση και με το opt-in για εκείνου οι οποίοι βρίσκονται σε χώρα άλλη αυτήν του δικαστή. Θα ήταν επίση σκόπιμο να υιοθετηθεί ένα opt-out για τα μικρότερα κατακεφαλήν ποσά ή ένα opt και ένα opt-in για τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ποσά και πάλι θα πρέπει να έχει όμως έναν οδηγό που θα παρακολουθεί ο δικαστής για να λάβει την απόφασή του. Υπάρχουν και άλλες λύσεις όπως αυτές του, του Αμερικανικού συστήματος που αποτελεί ένα είδος δεδικασμένου γενικού για τις διαφορές που έχουν ήδη κριθεί και θα μπορούσε να απαλλάξει τα κράτη από την υποχρέωση του opt-out επίσης, επιτρέψτε μας ε, να επιμείνουμε λίγο στα εργαλεία. Η οδηγία οπωσδήποτε θα ήταν ένα σημαντικό βήμα. Ωστόσο, στην επιλογή του νομοθετήματο. Ξέρουμε ότι και ο κανονισμό με την προστασία των δεδομένων μας έχει, που μα έχει οδηγήσει σε μελέτε για την ε, αξιολόγηση των υβριδικών κανονισμών αποδεικνύεται ότι θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο και αποτελεσματικό. Υπάρχουν όμω και κανόνε και πρόνοιε που δεν έχει καλύψει η πρόταση. Μεταξύ αυτών θα αναφέρω τις προϋποθέσεις παραδεκτού για την αγωγή αποκατάστασης, ε, το ομοιογενές των απαιτήσεων που προβλέπονται από τα προστατικά μέλη αυτή τη στιγμή, μητρό συλλογικής δράσης που θεωρούμε απαραίτητο, συλλογικής ε, αγωγής, συγγνώμη, θεωρούμε απαραίτητο και θα μπορούσε να εγκαθιδρυθεί με βάση και την εμπειρία των μητρών για τις ε, διαγραμμικές διαφορές ε, σε καταναλωτικές υποθέσεις. Επίσης, ε, η εισαγωγή ενός ταμείου θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί ως πρόταση, δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην πρόταση οδηγίας, αλλά και άλλες πρόνοιες απαγόρευση παραδείγματι ποσοστών επί του επιδικαστέτους ποσού. Για δε τις διασυνοριακές αγωγές παραδίδω το λόγο στη συνάδελφο. Σε ό,τι αφορά τις διασυνοριακές αγωγές, η σημερινή πρόταση έχει πολλά κενά. Ε, καθώς ε, η νέα αγορά πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο διασυνοριακών παραβάσεων. Οι ευρωπαϊκές αρχές το γνωρίζουν ε, γιατί έχουν αρχίσει να δίνουν μια απάντηση σε αυτόν τον πολλαπλασιασμό ε, των ε, διασυνοριακών κινδύνων ε, με τον κανονισμό του προηγούμενου Δεκεμβρίου που θεσπίζει μια συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμοδίες για την προστασία των καταναλωτών. Όμως, σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές αγωγές, τίποτα δεν προβλέπεται για να επιτρέψει στους ιδιώτες ή ε, επιχειρήσεις για άτομα να αναλάβουν άμεση δράση κατά μιας παράβασης ή για να λάβουν ηθική βλάβη. Ε, τώρα, η μελέτη παρουσιάζει διάφορα σημεία εμπλοκή. Παραδείγματο χάρη μα δείχνει ότι ο μηχανισμό εκπροσώπηση δεν είναι σαφής. Σήμερα μπορούμε να αναρωτηθούμε αν μια Βελγική Ένωση Καταναλωτών έχει τη δυνατότητα να δράσει για να εκπροσωπήσει καταναλωτές που ζουν στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Η μελέτη επιμένει επίσης για την δυσκολία σε ό,τι αφορά την ε, ε, τη δικαστική τη δικαιοδοσία. Παραδείγματο χάρη, το δικαστήριο που προστατεύει τον καταναλωτή ε, δεν είναι διαθέσιμο για τις συλλογικέ αγωγές. Σήμερα υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος πολλαπλασιασμού των συλλογικών αγωγών ε, με μία ε, Βελγική Ένωση που θα δρούσε ε, ε, για το, στο όνομα των Βέλγων καταναλωτών έναντι μιας εταιρεία που έχει έδρα στο Βέλγιο, μιας γερμανικής ένωσης που θα αναλάμβανε δράση στη Γερμανία. Έτσι λοιπόν μπορεί να έχουμε παράλληλες διαδικασίες χωρίς να μπορεί να υπάρχει συντονισμός των διαδικασιών αυτών. Βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα κάτι τέτοιο στην περίπτωση του Dieselgate, γιατί ξεπερνά τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόθεση αυτή. Έχουμε διαφορετικά μέρη κάθε φορά γιατί οι ενώσεις ε, που προσφέρουν στη δικαιοσύνη δεν είναι οι ίδιες. Έτσι λοιπόν διαπιστώνουμε ότι διαφέρουν τα μέρη και αυτό εμποδίζει να λειτουργήσουν οι μηχανισμοί του lease pendants που θα ήταν απαραίτητο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ στο γράφημα που δεν είναι και εξαντλητικό είχαμε αγωγές σε διάφορες χώρες, σε διάφορα δικαστήρια προσέφηγαν και καμία από αυτές τις αγωγές δεν είναι συντονισμένη. Υπάρχει όμως η λύση. Η πρώτη λύση θα συνιστατώ να πούμε ότι καθώς είμαστε σε μια ενιαία αγορά θα χρειαζόταν και μια ενιαία διαδικασία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα φιλόδοξη λύση, όμως αναμφισβήτητα είναι μια λύση που θα ανταποκρινόταν καλύτερα στην ιδέα της καλύτερης απονομής της δικαιοσύνης. Μία ισχυρή συνεργασία θα χρειαζόταν ε, για να ε, συσταθεί η υπόθεση και για να καθοριστεί η καλύτερη δικαιοδοσία που θα γνωρίζει καλύτερα την υπόθεση. Παραδείγματο χάρη, σε ό,τι αφορά στην εφραγκιότητα, προτείνουμε να χρησιμοποιήσουμε το κριτήριο ε, το κέντρο των κυρίων συμφερόντων, όμως εδώ θα αναφερόμαστε στα κύρια συμφέροντα της ομάδας των θυμάτων στην περίπτωση αυτή. Το ενδιαφέρον μιας νέας αγωγής θα ήταν ότι τελικά θα είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε μία και μόνο απόφαση για όλα τα θύματα, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους. Η πρόταση αυτή όμως προσκρούει σε ένα μεγάλο εμπόδιο του εφαρμοστέου δικαίου. Αν είναι μία η διαδικασία, προφανώς δεν θα υπήρχε παρά ένα εφαρμοστέο δίκαιο. Ε, ίσως να μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο στην περίπτωση δεν είναι πολλέ ακόμα, αλλά υπάρχουν στις περιπτώσεις όπου έχουν εναρμονιστεί οι νομοθεσίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. το χάρη μιλάμε για το δίκαιο των καταναλωτών και το ίδιο ισχύει και για την προστασία των δεδομένων. Μία δεύτερη λύση θα συνίστατο στο να ξεκινήσουν πολλές διαδικασίες, ε, πολλές προσφυγές στη δικαιοσύνη, όμως να είναι συντονισμένες. Υπάρχει ήδη λύση στον τομέα της αφαιρεγγιότητας, και υπάρχει επίσης το τομέα της προστασίας των δεδομένων, όμως εδώ δεν μιλάμε ε, για ε, διαδικασίες δικαιοδοτικές, αλλά ουσιαστικά ε, μιλάμε για διαδικασίες που υλοποιούνται από τις αρχές προστασίας των δεδομένων. Και υπάρχει και μια συντονισμένη διαδικασία που έχει προβλεφθεί από τον κανονισμό του Δεκεμβρίου 2017 για τις αρχές που για την προστασία των καταναλωτών. Έχουμε λοιπόν μια κύρια διαδικασία και δευτερεύουσες διαδικασίες. Σύμφωνα με το γράφημα που βλέπετε εδώ, αυτό προποθέτει μια πραγματική συνεργασία των δικαιοδοσιών και πραγματική διαδικασία των διαδικασ... πραγματικό συντονισμό των διαδικασιών. Όμως είναι δυνατόν και αυτό. Οι λύσεις 1 και 2 μπορούν να είναι σωρευτικές, όπως συμβαίνει σε ό,τι αφορά ε, την αφαιρεγγιότητα, όπου έχουμε μια συλλογική διάσταση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία, οι συνάδελφοι έχουν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις και στις δύο προσκεκλημένες. Κύριος Λεμπρετών. Ευχαριστώ. Τις ε, δύο ο που μας παρουσίασαν με πολύ ενδιαφέρουσε παρατηρήσεις του και χαίρομαι πολύ που ξαναβλέπω την κυρία Ζώ την έχω γνωρίσει σε άλλο βήμα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις Βρυξέλλε. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτές τις συλλογικέ αγωγές, είναι πράγματι ένα πραγματικό πρόβλημα. Υπάρχουν όλο και περισσότερε διασυνοριακέ παρεμβάσει στο καταναλωτικό δίκαιο αυτό που πρέπει να αποφύγουμε ένα και μόνο διασυνοριακό αδίκημα ε, να είναι αντικείμενο ε, διαφορετικών αγωγών ε, σε εθνικά δικαστήρια. Είναι κάπως παράλογο αν το δούμε αυτό από τη σκόπια των θυμάτων. Επομένως, ναι, γιατί να μην φανταστούμε ένα είδος εναρμόνισης, όμως προφανώς αυτό θα είναι δύσκολο. Τώρα, η βασική μου ερώτηση είναι για να αποφύγουμε ακριβώς αυτές τις παράλληλες συλλογικέ αγωγές όπως έχουμε στην περίπτωση του Dieselgate τι θα κάνουμε η κυρία Ζώ πρότεινε να δούμε που βρίσκονται τα κύρια συμφέροντα της ομάδας των θυμάτων δεν έχω κάποια αντιπρόταση όμως δεν σας φαίνεται ότι είναι δύσκολο να μαντέψουμε ποιο είναι το κέντρο των ε, κυρίων συμφερόντων ε, των θυμάτων. Ε, μιλήσουμε για το Τζελγκέιτ, νομίζω είναι η Γερμανία στην περίπτωση αυτή. Αλλά για να εμβαθύνουμε. Αν κατάλαβα καλά και αν είναι η Γερμανία, τότε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ασκηθεί μια συλλογική αγωγή στη Γερμανία, εφαρμόζοντας το γερμανικό δίκαιο λοιπόν θέτει προβλήματα αυτό, όπως έχουν τα πράγματα σήμερα. Μήπως ε, θα πηγαίναμε προς μια μεγάλη, πολύ μεγάλη εναρμόνιση. Δηλαδή το πλεονέκτημα στην Επιτροπή αυτή είναι ότι <laughs> είναι ε, τα νομικά προβλήματα που ε, έρχονται το ένα μετά το άλλο και γενικά για να τα επιλύσουμε προτείνουμε πάντοτε μία εναρμόνιση. Παραδείγματο χάρη προτείναμε προλίγου ένα ευρωπαϊκό εμπορικό δικαστήριο και πολύ σύντομα ίσως να έχουμε μια εναρμονιση το χαρη προτειναμε προλιγου ενα ευρωπαικο Αρχή Εργασίας. Το πρόβλημα είναι, in fine, έχουμε μία τάση να περιθωριοποιούμε όλο και περισσότερο το εθνικό δίκαιο έτσι λοιπόν, ε, να σας ρωτήσω, δεν φοβάστε ότι αυτή η εναρμόνιση που φαίνεται επιθυμητή όταν σκεφτόμαστε έτσι φυρημένα, μήπως κινδυνεύσει να καταλήξει σε περιθωριοποίηση υπερβολική των εθνικών διαδικασιών. Παρακαλώ, κύριος Βόλκιν. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω ρωτήσω πολύ τις προσεκλημένες για την παρουσίαση της μελέτης. Ε, νομίζω πως ε, παρουσιάζονται ορισμένε πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές στη μελέτη αυτή. Ε, μόνο αν διαβάσει κανείς την περίληψη μαθαίνει πολλά. Αναφέρεται δηλαδή εκεί ότι το υφιστάμενο σύστημα, και διαβάζω, δεν είναι επαρκές και πως χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μία νέα πρόταση για όλους αυτούς τους λόγους που εκθέσατε. Από την άλλη, η... Από τη μία, η, μία, η πρόταση αυτή πρέπει να διασφαλίζει πρόσβαση, από την άλλη θεωρώ πάρα πολύ καλό ότι το πεδίο εφαρμογής, το οποίο ε, προτείνεται, είναι πολύ στενό. και, δεν πρέπει, και περιορίζεται σε συγκεκριμένες ε, μορφές, ενώ θα έπρεπε να επεκταθεί, να διευρυνθεί και να αφορά και άλλα νομικά πρόσωπα. Όλα αυτά δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή νομικά δεν είμαστε ικανοποιημένοι, τα πράγματα δεν είναι όπως τα θέλαμε και τα παραθύματα που αναφέρατε ήταν πάρα πολύ καλά. Στη συζήτηση αναφέρθηκαν ορισμένες πληροφορίες τις οποίες ε, θεωρώ πως, τις οποίες θεωρώ ε, μη ισορροπημένες. Νομίζω πως ορισμένες είναι λανθασμένες μάλιστα. Θεωρείται ότι μία διεύρυνση της νομικής προστασίας θα ε, οδηγήσει σε μια βιομηχανία αγωγών όπως αυτό που βλέπουμε στις Ηνωμένε Πολιτείες. Όλες οι χώρες ε, που εξετάσατε δεν κινδυνεύουν να γίνουν ακριβώς ε, όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε, να δημιουργηθεί βιομηχανία αγωγών. Μετά, πιστεύω πως ε, πολύ σωστά καταστήσατε σαφές στη σελίδα 65 ότι έχουμε ανάγκη ενός δεσμευτικού μέσου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφερθήκατε επίση στο πεδίο εφαρμογή, το είπα ήδη πως πρέπει να διευρυνθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει και τα φυσικά πρόσωπα. Μπορείτε να μας πείτε γιατί είναι τόσο σημαντικό για σας ε, να συμπεριλαμβάνονται και τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα και όχι μόνο ενώσεις. Το άρθρο 4 παράγραφος 4 μπορεί να αποβεί αρκετά επικίνδυνο. Θα θέλαμε λοιπόν περισσότερες διευκρινήσεις γι' αυτό. Τι εννοείται. Επίσης να πω πως ε, φοβάμαι ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων δεν θα εξετάσει περισσότερο την πρόταση του ΙΣΥ για αυτό, δηλαδή που αναφέρετε κι εσείς ότι θα γίνει, τι χρειάζεται η Ευρώπη και πως οι καθυστερήσεις θα αποβούν επιζήμιες. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις και να σας ζητήσω να απαντήσετε, αλλά σας παρακαλώ σύντομα. Θα απαντήσω στην ερώτηση που τέθηκε από τον κύριο Λεμπρετών και εγώ τον χαιρετίζω. Πραγματικά βάλατε το, το δάχτυλο στην πληγή στο πρόβλημα που έχει να κάνει με το κριτήριο των αρμοδιοτήτων, το αναφερθήκαμε στο κέντρο των συμφερόντων της ομάδας των θυμάτων. Στο Dieselgate είναι πράγματι δύσκολο να φανταστούμε που βρίσκεται αυτό το κέντρο των κοινών συμφερόντων των θυμάτων και αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στο να προτείνουμε, παραδείγματο χάρη, ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση στα γερμανικά δικαστήρια όπου είναι το δικαστήριο των εναγωμένων. Και όμως ίσως σε άλλες περιπτώσεις να μην ανταποκρίνεται ε, το δικαστήριο ε, του εναγωμένου σε ένα νέο σύστημα ίσως θα έπρεπε να έχουμε μία συνεργασία για να καθορίσουμε ποιος είναι ο αρμόδιος δικαστής. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κίνδυνο υπερβολικής εναρμόνισης από τη στιγμή που ξεκάθαρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως σε ό,τι αφορά το καταναλωτικό δίκαιο, έχουμε ένα ε, δίκαιο προστασίας που είναι όλο ένα και πιο ισότιμο στα διάφορα κράτη-μέλη. Τώρα στο να προβούμε σε εναρμόνιση των υλικών κανόνων μέσω της εναρμόνισης των δικονομικών κανόνων δεν ε, είναι μια φιλοδοξία εντελώς ασύμετρη. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές. Ε, μας δίνουν την ευκαιρία να είμαστε πιο συγκεκριμένες. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα με την δυνατότητα να δημιουργηθεί μια βιομηχανία συλλογικών αγωγών. Φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές ε, δικλείδες ασφαλείας που έχουν ληφθεί για να αποφευχθεί μια τέτοια βιομηχανία. Και μια αρχική παρατήρηση στη χώρα που αναπτύχθηκε τέτοια βιομηχανία έγινε για άλλους λόγους πέρα από τους μηχανισμούς συλλογικής προσφυγής στις Ηνωμένες ε, ε, Πολιτείες. Ε, έχουμε ένα λαϊκό δικαστή, ενώ εδώ έχουμε ένα νομικό δικαστή. Επίσης, αποκλείονται εντελώς οι αποζημιώσεις για ηθική βλάβη και δεν φαίνεται τα κρατημέλη να είναι έτοιμα. Αναφέρω το άρθρο 6 που έχουν περιορίσει την επανόρθωση που μπορεί να δοθεί. Υπάρχει το contingency fees, ε, παραδείγματο χάρη, τα οποία συνεισφέρουν ε, στο να θεωρούνται οι συλλογικές αγωγές ε, κάτι που ευνοεί τους δικηγόρους και όχι την ομάδα των θυμάτων. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε σήμερα τέτοιο κίνδυνο να δημιουργηθεί βιομηχανία αγωγών στην Ευρώπη, γιατί είναι δεσμευτικό μέσο. Αυτό σχετίζεται με το τελευταίο θέμα, με τις ε, επιπτώσεις. Γιατί δεσμευτικό μέσο. Γιατί σήμερα βλέπουμε ότι είναι άνηση η κατάσταση και αν αναπτυχθεί η εσωτερική αγορά θα πρέπει να αναπτυχθεί και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αγορά αυτή. Σήμερα δεν ισχύει. Δηλαδή, Όπου και να είσαι πρέπει να προστατεύεσαι, όπου και να βρίσκεται ο καταναλωτές, το δίκαιο θα πρέπει να είναι το ίδιο και θα πρέπει να έχει εναρμονισμένα εργαλεία λοιπόν. Εξού και το θέμα της ε, συμμετοχής ε, σήμερα τη συμμετοχή τη κοινωνία. Αν ε, δώσουμε στην κοινωνία ένα εργαλείο με αυτέ τι ασφαλιστικέ δικλείδε, είμαστε στη σωστή οδό. Γιατί για, μιλάμε για νομικά πρόσωπα. Εδώ προτείνουμε να υπάρχουν νομικά πρόσωπα που να μπορούν να είναι μέλη της ε, ομάδας ε, των ε, εναγόντων. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο, παραδείγματο χάρη, να γίνει διάκριση σε ορισμένες περιπτώσεις μεταξύ των καταναλωτών, τελικών πελατών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν μιλάμε περισσότερο για την σύλληψη της ομάδας ε, και μπορεί αυτά τα φυσικά άτομα να εντάσσονται στην κατηγορία των καταναλωτών. Τώρα για το άρθρο 44, συγγνώμη 84, δεν ε, αποτελεί κίνδυνο. Αυτό που σας ε, έδειξα στις διαφάνειες ε, που χρειάζονται βελτιώσεις. Αυτό συνδέεται με τη δυνατότητα που δίνεται στα κράτη-μέλη να περιορίσουν ε, ουσιαστικά τα ένδικα μέσα που μπορεί να αναζητήσουν τα άτομα που έχουν ενεργητική νομιμοποίηση. Δηλαδή, μπορεί, παραδείγματο χάρη, τα άτομα να αναζητήσουν να προσφύγουν σε κάποιε χώρε, ε, εκεί όπου μπορούν να λάβουν αποζημίωση και να αποφύγουν κάποιε άλλε χώρε όπου δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις ε, δύο προσκεκλημένες. Φυσικά και είστε πρόσδεκτε να παραμείνετε στην αίθουσα για την επόμενη ακρόαση που έχει το ίδιο θέμα, τη συλλογική προσφυγή και την βελτιωμένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους, με ερωτηματικό. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους ομιλητές μας λοιπόν για την ακρόαση αυτή, την καθηγήτρια Σουζάννα Αουγγενχόφερ, καθηγήτρια αστικού δικαίου, ευρωπαϊκού ιδιωτικού δικαίου, συγκριτικού δικαίου και ε, ρύθμιση της αγορά, και δικαίου ρύθμιση αγοράς μέσω καταναλωτικού δικαίου και δικαίου του ανταγωνισμού στο Πανεπιστημίο Humboldt του Βερολίνου και τους Λόρα Μάρκους και Σίμον Νοβέμπερ από την Ένωση Καταναλωτών του Βελγίου Τεστ Ασάμ. Καθηγήτρια Ούγκενχόφερ. συμμετείχατε στην κατάρτιση της γερμανικής νομοθεσίας για τις συλλογικέ αγωγές και σας ζητήσαμε μια αξιολόγηση της πρότασης οδηγίας από την οπτική γωνία του ερευνητή. Ο, η κυρία Μάρκους και ο κύριος ε, Νοβέμπερ από το Βέλγιο είναι εδώ, ότι το Βέλγιο έχει μία από τις πιο αναπτυγμένες νομοθεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα συλλογικής αγωγής και η Ένωσή σας έχει συμμετάσχει σε πολλές τέτοιες ε, περιπτώσεις συλλογικών αγωγών. Θα μοιραστείτε λοιπόν την εμπειρία σας μαζί μας. Οι προσκεκλημένοι έχουν κληθεί να απαντήσουν στο ακόλουθο ερώτημα. Καταρχάς, υπάρχουν δικονομικές εγγυήσεις για την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που να είναι τόσο κατάλληλες και επαρκείς έτσι ώστε να ε, αποφεύγονται οι περιπτώσεις ε, κατάχρησης. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω πρώτα το λόγο στην καθηγήτρια Άουγκενχόφερ για 10 λεπτά και μετά στην κυρία Μάρκους και τον κύριο Νοβέμπερ για άλλα 10 λεπτά για τις παρουσιάσεις τους και έπειτα τα μέλη της Επιτροπής θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις. Κύριε Όγκενχόφερ, έχετε το λόγο και 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Και μια που έχω μόνο 10 λεπτά στη διάθεσή μου, θα εστιάσω μόνο σε ορισμένα σημεία. Ας αρχίσουμε από τα καλά νέα. αισθάνομαι μεγάλη ανακούφιση για το ότι έχουμε επιτέλους μία πρόταση. Πολλοί από εσά και εγώ χάρηκαν όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη πως ε, είναι δυνατόν να ζητήσει κανείς αποζημίωση σε περίπτωση παραβίασης ε, της νομοθεσίας και υπάρχει δυνατότητα λοιπόν ε, για συλλογικές αγωγές. Θεωρώ επίσης ότι το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου καταλληλότητας του fitness check του καταναλωτικού δικαίου της ε, Ένωσης έδειξε πως μία από τις μεγαλύτερες ελλείψεις, σημαντικότερες ελλείψεις του καταναλωτικού δικαίου είναι η έλλειψη μηχανισμών επιβολής. Ήδη το 2015 υπάρχουν αναφορές για διάφορες τέτοιες ε, περιπτώσεις ανεπιτυχούς και ανεπαρκούς εφαρμογής και επιβολής της νομοθεσίας. Πολλές από αυτές έχουν χαρακτηριστεί ως fake news. Η, περίπτωση της υπόθεσης της ε, Volkswagen που έλαβε φυσικά πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις αποδεικνύει ότι η έλλειψη συλλογικής αγωγής είναι μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη και στη Γερμανία η οποία βέβαια πρόσφατα θέσπισε ένα σύστημα συλλογική εισαγωγή, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου. Βέβαια δεν είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Η διαδικασία όμως ε, αυτή η πρόταση παρέχει τη δυνατότητα μιας διαδικασίας σε ένα στάδιο. Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις αυτή τη στιγμή που εκδικάζονται στην ε, Γερμανία, στις οποίες συμμετέχουν ε, συλλογικά. Το κόστος επίσης είναι πολύ απαγορευτικό για έναν μεμονωμένο καταναλωτή. Το γερμανικό δίκαιο δεν απαγορεύει στους καταναλωτές να προσφύγουν στο δικαστήριο, όμως ακριβώς επειδή το κόστος είναι τόσο απαγορευτικό και τα ένδικα μέσα πρέπει, έχει θεσπιστεί αυτή η νομοθεσία για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτές οι εξελίξεις είναι θετικές και αυτό αναφέρεται και στην πρόταση. Μετά, το επόμενο θετικό είναι ότι η γερμανική νομοθεσία ακριβώς ε, προβλέπει μια διαδικασία σε ένα στάδιο και αν είστε γερμανός πολίτης ή βρίσκεστε στη χώρα και μιλήσετε με ε, άτομα που είναι υπέρ αυτής της αναγνωριστικής αγωγής αυτών των προτύπων Musterfest Stellungsklage στα γερμανικά θα δείτε ότι με τη θέση σε ισχύ του νόμου υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Στην περίπτωση της Volkswagen, για παράδειγμα, όλοι οι καταναλωτές, όσοι δηλαδή είχαν αγοράσει αυτοκίνητα Volkswagen και δεν είχαν τα οικονομικά μέσα για να προσφύγουν, θα καταφέρουν επιτέλους να δικαιωθούν. εκπρόσωποι ενώσεων καταναλωτών, μάλλον οι όσοι συμμετέχουν σε ενώσεις καταναλωτών δεν θα, έχουν ε, την, δεν, θα, δεν θα είναι υποχρεωμένοι να προσλάβουν δικηγόρο. Βέβαια, αν επισκεφτεί κανείς τον ιστότοπο της Ένωσης Καταναλωτών και δει τις ε, συχνές ερωτήσεις, θα δει πως ε, υπάρχουν αναφορές στην περίπτωση της ε, Volkswagen, του σκανδάλου με Dieselgate. Εκεί αναφέρεται ότι οι καταναλωτές με μεμονωμένοι καταναλωτές πρέπει να συμβουλευτούν δικηγόρο και να ζητήσουν νομική συμβουλή έτσι ώστε να κάνουν όλες τις κατάλληλες ενέργειες. Είναι λοιπόν μια καλή περίπτωση, όμως δεν θα πρέπει να είναι πανάκια ε, και το μόνο πράγμα που θα, από το οποίο θα δηλήσει έμπνευση η Επιτροπή όταν θα καταρτήσει την πρόταση. Τώρα, άρθρο 6.3β. Εδώ αναφέρονται οι μικρές αγωγές, οι, διαφορές, οι αγωγές για διαφορές μικρής αξίας, όπου υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι της ε, γερμανικής νομοθεσίας εδώ στην πρόταση της Επιτροπής. Οι μονομένοι καταναλωτές θα έχουν τη, την δυνατότητα να ε, λαμβάνουν τις αποζημιώσεις. Τώρα, ποια είναι τα αρνητικά. Σε γενικές γραμμές, η πρόταση σε πολλά σημεία είναι υπερβολικά ασαφής. Παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα λοιπόν, στην επόμενη διαφάνεια, είναι ότι υπάρχει δυνατότητα υποβολής αγωγής σε περίπτωση που βλάπτονται τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών. Συλλογικά συμφέροντα ενό αριθμού καταναλωτών. Ποιο είναι όμως το σωστό νούμερο, σωστός αριθμός είναι ένα, είναι 20, είναι παραπάνω. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ασάφεια και εάν η περίπτωση αυτή, εάν η πρόταση αυτή εγκριθεί, τότε θα είναι αρμόδια τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν ποιο θα είναι ο ρυθμό. Ε, η Γερμανία, α πούμε, μπορεί να αποφασίσει ότι τρει ε, καταναλωτέ αρκούν. Η Ιταλία μπορεί να επιλέξει άλλον αριθμό. Αυτό είναι ει βάρο των καταναλωτών αλλά και των επιχειρήσεων. Μετά, το άρθρο 4, παράγραφος 4. Τον έφεραν οι συνάδελφοι. Εδώ πιστεύω υπάρχει κίνδυνος να γίνει κατάχρηση από τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένε οντότητες. Μπορεί να υπάρχει απροθυμία ε, συλλογική εισαγωγή. Στη Γερμανία έχει συμβεί αυτό με την χρήση αυτή της, ε, των προτύπων αγωγής. Υπάρχει τόσο στενό πεδίο εφαρμογής ε, με αυτήν την νομοθεσία που εγκρίθηκε στη Γερμανία, ώστε μόνο μία ένωση καταναλωτών ε, είναι σε θέση να καταθέσει τέτοια αγωγή. Επίσης υπάρχουν προβλήματα οικονομικού χαρακτήρα. Το άρθρο 15.1 επίσης αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα ε, για να επιτρέψουν σε εγκεκριμένες οντότητες να καταθέτουν αγωγές. Όμως, και εδώ υπάρχει μεγάλη ασάφεια, πράγματι θα μειωθεί το κόστος ε, των ε, δικαστικών διαδικασιών, όμως εδώ δεν ε, μας εγγυάται η πρόταση ασφάλεια δικαίου. Μετά, σε περιπτώσεις καταχρήσης, εδώ δεν βλέπω κίνδυνο να εισβάλλουν αμερικανικές ε, νομικές εταιρείες στην ε, αγορά, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο το κέρδος. Θα έλεγα πως αυτό που με ενοχλεί στην πρόταση είναι η σχέση ανάμεσα στις μεμονωμένες αγωγές και στις ε, συλλογικές αγωγές. Οι συνάδελφοι ήδη είπαν ότι το άρθρο 6 είναι αρκετά ασαφές και διαβάζοντας το αρκετές φορές κατάλαβα, δεν ξέρω, μπορεί να φταίω εγώ, μπορεί εγώ να μην είμαι αρκετά <laughs> μορφωμένη, αλλά έπρεπε να το διαβάσω πολλές φορές για να καταλάβω ότι σύμφωνα με το άρθρο 10, μία απόφαση μπορεί να έχει επιπτώσει σε όλους τους καταναλωτές. Το άρθρο 10 λέει ότι μία απόφαση είναι δεσμευτική για όλους. Επίσης, η πρόταση έχει αρνητικέ επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, το, στο άρθρο 10 λέει ότι η απόφαση θα είναι δεσμευτική μόνο αν είναι υπέρ του καταναλωτή. Στην περίπτωση αυτή η γερμανική νομοθεσία είναι καταλληλότερη και είναι πάντα δεσμευτική για τον καταναλωτή ο οποίος αποφασίζει να εισέλθει σε μια τέτοια διαδικασία. Η απόφαση θα πρέπει να είναι δεσμευτική έτσι κι αλλιώς. Τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω υπάρχουν κάποιες ε, διαρθρωτικές αλλαγές που προτείνω. Δηλαδή, γιατί να μην πάμε ένα βήμα παραπέρα και να επιτρέπουμε στους καταναλωτές να συμμετέχουν ως μια οντότητα. Ιδανικά βέβαια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση στη συλλογική αγωγή. Προσωπικά είμαι υπέρ ε, της ευελιξίας έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται τροποποιήσεις στον ε, κανονισμό ως προς το ποιες παραβιάσεις θα ενεργοποιούν την εφαρμογή της οδηγίας. Τώρα, δεν νομίζω πως ε, η πρόταση είναι χάλια τελείως, νομίζω πως η προσέγγιση Επιδέχεται κάποιες αλλαγές, ίσως τις χρειάζεται κιόλα. Και νομίζω πως δεν θα πεθάνει και κανείς αν καθυστερήσει λιγάκι. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ, Μάρκους και Νοβέμπερ, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Έχετε μήπως το τηλεχειριστήριο για τις διαφάνειες. Um, Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας μιλήσουμε για τον ε, Ευρωπαϊκό, για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για Συλλογική Αγωγή που μας κάνει όλους πολύ περήφανος, ώρα που ξέρουμε επίσης ότι έχει και τις αδυναμίες του και τα τις ελλείψεις του. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί έχω πολύ λίγο χρόνο. Θα περάσω έτσι γρήγορα γρήγορα τις πρώτες ε, διαφάνειες. Είμαστε η Τεστασά, είμαστε η μεγαλύτερη Ένωση Καταναλωτών του Βελγίου με 300.000 μέλη. Εχθές ε, γιορτάσαμε την 60η επέτειο από την ίδρυσή μας και πάνω από όλα είμαστε απόλυτος ανεξάρτητοι. Δεν υπάρχει ούτε διαφήμιση, ούτε επιδότηση, ούτε άλλη οικονομική ε, βοήθεια. Ο νόμος λοιπόν για την συλλογική αγωγή του Βελγίου 2014. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι δύσκολο για τον καταναλωτή να καταφύγει στα δικαστήρια και πολύ συχνά δεν μπορεί και να βρει το δίκαιο του. και στην επόμενη διαφάνεια, ε, για να περιγράψω ότι αρχικά είχε σχεδιαστεί μόνο για εμπορικές διαφορές αυτός ο ε, νόμος, τώρα απευθύνεται και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχει να κάνει με ζημία που προκύπτει μετά την 1η Ενάτου του 2014 με ρητή αναφορά 31 νομοθετημάτων είτε ευρωπαϊκών είτε βελγικών που εάν παραβιαστούν εφαρμόζεται ο νόμος για την ε, συλλογική αγωγή. Αφήνω στην άκρη το διάγραμμα την αρχιτεκτονική του νόμου και προχωρώ ακόμη περισσότερο για να φτάσω εδώ στην σύνοψη της εφαρμογής. Πρώτα λοιπόν πρέπει να γίνει η αίτηση ενώπιον του δικαστή για να κρυθεί το παραδεκτό και να ανοίξει η διαδικασία opt-in, opt-out. Ως προς την κρίση του παραδεκτού εξετάζει ο δικαστής εάν είναι επαρκή αντιπροσωπευτική η αγωγή. Δεύτερον, εάν υπάρχει παραβίαση είτε συμβατική είτε εξωσυμβατικής ε, ρήτρα, δηλαδή κάποιε νομοθεσίε από τις 3, τα 31 νομοθετήματα που αναφέρονται. Και αν υπάρχει τρίτον, ε, καλύτερο τρόπο αποκατάσταση των δικαιωμάτων των καταναλωτών από αυτών τη συλλογική αγωγή. Και άπαξ και αποφασίσει για το παραδεκτό ο δικαστή, ορίζει και πάμε πίσω στο σχεδιάγραμμα, ορίζει εάν θα ε, προχωρήσει με την επιλογή του opt-in ή του opt-out. Μετά την ε, φάση αυτή να αρχίζουν υποχρεωτικές ε, διαβουλεύσεις, υποχρεωτικές για την επιτεύξη συμφωνίας, εξοδικαστικής δηλαδή, που πάντα όμως είναι δυνατή είτε πριν από την κατάθεση της αγωγής, κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής συνδιαλλαγή, είτε και ε, στη φάση όπου έχει αποφασίσει επί τη ουσία τη απόφαση ο δικαστή. Μετά λοιπόν τι υποχρεωτικέ αυτέ διαβουλευσει μπορεί να προκύψει όπω είπα ε, συμφωνία των μερών εξοδικαστική την οποία, την οποία εγκρίνει ο ε, δικαστής και ορίζει διαιτητή ή εν αρμόδιο για την διευθέτηση αυτή τη διαφορά εξοδικαστικά και αν αυτό δεν επιτύχει τότε θα πρέπει να κρίνει ο ίδιο ο δικαστή την ουσία τη υπόθεση. Ε, και θα προχωρήσω για να μιλήσω για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της νομοθεσίας μας. Βεβαίως δίνει μια φωνή στον καταναλωτή αυτό το νομοθέτημα. Τους επιτρέπει δηλαδή να προσφύγουν στα δικαστήρια για δικαιώματα τους που διαφορετικά θα μπορούσαν να διεκδικήσουν και αποτέλεσε ισχυρό μέσο πίεση. Ένα παράδειγμα, το 2015 ξεκινήσαμε μια αγωγή κατά της εταιρεία της αεροπορικής της Thomas Cook για μια υπόθεση οκτάωρης καθυστέρησης πτήσης από την Τενερίφη στις Βρυξέλλες η οποία οφειλόταν σε μια σύγκρουση αεροσκαφών πάνω στον διάδρομο αποκείωσης, την οποία είχε επικαλυστεί ω ανωτέρα βία η Thomas Κουκ και δεν ήθελε να ε, προσφέρει την αποζημίωση που προβλέπεται από τον κανονισμό 2004 για του επιβάτε σε περίπτωση καθυστέρηση. Εμείς, ε, αφού μπορέσαμε να, συλλέξουμε αρκετούς, να συγκεντρώσουμε αρκετού ενδιαφερόμενου καταναλωτέ και να ξεκινήσουμε αυτή την ε, διαδικασία, χωρί να περιμένουν καν τη διαδικασία παραδεκτού από το δικαστή η Thomas Cook αποζημίωσε. Και άρα θέλω να υπογραμμίσω ότι μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό μέσο πίεσης μια τέτοια συλλογική αγωγή. Ταυτόχρονα επισημαίνω ότι για 400 ευρώ κανένα καταναλωτή μόνο δεν θα κατεφεύγει στα δικαστήρια, γιατί είναι πολύ ακριβά τα. Οι αμοιβέ είναι πολύ ψηλέ οι αμοιβέ των δικηγόρων και όλη η διαδικασία πολύ ακριβή. Ε, εξού και αποδείχθηκε πολύ χρήσιμη αυτή η δυνατότητα για συλλογική αγωγή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στην επόμενη διαφάνεια επίση υπάρχουν και μειονεκτήματα βέβαια, καταρχά γιατί είναι χρονοβόρα η διαδικασία όπω την προβλέπει ο νόμο και ότι δεν ήταν πρόθεση του ε, όνο του νομοθέτη να γίνεται μια διαδικασία χωριστή ε, για, το παραδεκτό, επειδή ακριβώς ε, διαρκώς γίνονται στάσεις παραδεκτού και υπάρχουν και άλλα ζητήματα που με την ευκαιρία αυτή εισάγονται, επί της ουσίας δηλαδή, περνάει πολύ καιρό άπαξ και, και οριστεί ότι είναι παραδεκτή η αγωγή, μπορεί κανείς να κάνει προσφυγή ή μάλλον αγωγή, μάλλον έφεση κατά της απόφασης περί παραδεκτού και αυτό βέβαια οδηγεί σε ακόμη μακρύτερες ε, διαδικασίες. Ε, ένα άλλο παράδειγμα που μπορώ να σας προσφέρω ήταν ε, η επαναπόληση εισιτηρίων για συναυλία σε υπέρογκα, με υπέρογκα ποσά. Ξεκινήσαμε τη σχετική διαδικασία το 2014 και είχαμε την προηγούμενη μόλις εβδομάδα την δικάσιμο για την παρουσίαση των θέσεων των διαδίκων όπως είπα για τα δικά μας ζητήματα και μια από τις ακόμη αδυναμίες του ε, νόμου αυτού είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να κερδίσουμε κάποια αμοιβή, δεν υπάρχουν εργολαβικές δηλαδή δικηγορικές αμοιβέ που να προβλέπονται σε αυτήν την περίπτωση των συλλογικών αμοιβών, ακόμη και σε περίπτωση αποζημίωσης ε, και άρα ε, αυτό είναι άλλη μια αδυναμία της νομοθεσίας. Ένα άλλο σημείο είναι ότι καλύπτει η ζημία που έχει προκύψει μόνο την 1η του 2014. Για τη Volkswagen, παραδείγματι, μπορούμε να ε, εκπροσωπήσουμε καταναλωτές που έχουν αγοράσει ε, αυτοκίνητο με πειραγμένο λογισμικό για το θέμα των ε, εκπομπών μόνο εφόσον αυτοί το αγόρασαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2014 και εφαρμογή του νόμου. Οι προηγούμενοι δεν μπορούν να καλυφθούν από τη συλλογική αγωγή. Ε, Επίση, μια διαδικασία opt-out πολύ σημαντική είναι, κατά συγκαταλέγεται μεταξύ των αδυναμιών τη νομοθεσία. Υπήρχε μια απόφαση για opt-in για μεγάλο ε, μια μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών και έτσι υποχρεώθηκε αυτή να αποστείλει επιστολή σε κάθε καταναλωτή για να ε, ζητήσει να κάνουν το opt-in κτλ. Αλλά ήταν τόσο περίπλοκη η διαδικασία που δεν μπόρεσε κανένα καταναλωτή να την αντιληφθεί. Ή μάλλον η επιστολή, το κείμενο τόσο περίπλοκο που δεν μπόρεσε κανένα καταναλωτή να αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό και φυσικά και το έκανε επίτηδε ε, η εταιρεία αυτή των τηλεπικοινωνιών για να μην ε, κάνουν το opt-in οι καταναλωτέ, γιατί αυτό θα κόστησε πολύ περισσότερα χρήματα στην εταιρεία και νομίζω ότι αυτό πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό. Ευχαριστώ. Θα κάνω ένα σχόλιο για την πρόταση. Καταρχήν, το επίπεδο της εναρμόνισης. Ζητήσαμε ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης ε, για να διατηρηθεί η φυστάμενη διαδικασία γιατί περίπτωση χάρη η διαδικασία στο Βελγίο προστατεύει περισσότερο τους καταναλωτές. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα υιοθετήσουμε ένα άλλο σύστημα συλλογικών αγωγών ε, βάσει τη οδηγία. Ε, ε, αντί να διατηρήσουμε το δικό μα σύστημα. Δεν είναι λογικό αυτό. Θέλουμε λοιπόν ένα ελάχιστο επίπεδο εναρμόνιση που να μα επιτρέψει να διατηρήσουμε τη δική μα διαδικασία. Κατόπιν, συνδέουμε τη διαδικασία με τι αγωγέ επιπαραλήψη. Είναι δύο διαφορετικέ ε, διαδικασίε αυτέ. Πρέπει να γίνονται ανεξάρτητα, είναι χρονοβόρε και πολλές φορές ε, δεν χρειάζεται αγωγή παραλήψη γιατί έχει σταματήσει η ζημία σε σχέση με τις ε, δυσκολίες της προσωπικοποίησης των ζημιών. Ε, αναφέρθηκε η καθηγήτρια σε αυτό. Το άρθρο 6.2 προβλέπει δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να παρεκκλίνουν από την κύρια διαδικασία συλλογικών αγωγών και απλώς να υπάρχει μια δήλωση ευθύνης του εμπόρου και κατόπιν θα πρέπει ε, ο καταναλωτής ε, να προβεί σε δική του ατομική αγωγή. Αυτό δεν είναι το πνεύμα των συλλογικών Πρέπει να διαγραφεί αυτή η διάταξη, γιατί ποτέ δεν θα προσφύγει μόνο του καταναλωτή στο δικαστήριο. Στη Volkswagen, ε, παραδείγματο χάρη, το λεγόμενο Dieselgate, οι καταναλωτέ ε, είχαν αγοράσει αυτοκίνητα με διάφορε μηχανέ, με διάφορου κινητήρε τα είχαν χρησιμοποιήσει διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Ένα κράτο μέλο αποφασίσει εδώ να χρησιμοποιήσει την παρέκκληση στην πρόταση. Ο δικαστή θα αποφασίσει μόνο για την ευθύνη του εμπόρου, ότι τότε ο καταναλωτή θα πρέπει να ε, προβεί σε, συλλογή, σε αγωγή που θα πρέπει να αποδείξει το σύνδεσμο μεταξύ της ευθύνης ε, του εμπόρου Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη η πιθανότητα ότι ποτέ δεν θα γίνει μια τέτοια αγωγή σε ό,τι αφορά τι ε, υποθέσει όπου έχουμε χαμηλές ζημίες. Ακόμη και αν είναι μικρό το ποσό, τι σημαίνει μικρό ποσό. Παραδείγματο χάρη χρεώνει μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών 8 ευρώ παραπάνω. Σε κάποιο καταναλωτή αυτό θεωρείται μικρό ποσό. Και αν ε, υιοθετηθεί, θα πρέπει να συνδυαστεί με ένα σύστημα opt-out, διαφορετικά ο καταναλωτής ποτέ δεν θα πει θέλω να είμαι μέλος της ομάδας, αν δεν λάβω επανόρθωση και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα σχέδιο backup, παραδείγματο χάρη, όταν δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς ποιο είναι ο καταναλωτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των ε, υποθέσεων, έχουμε πολλές προτάσεις, παραδείγματο χάρη, οι ε, ζημίες, οι αποζημιώσεις, συγγνώμη, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ε, στην περίπτωση που θέλουμε να ξεκινήσουμε μία νέα συλλογική αγωγή για τη χρηματοδότηση του τρίτου μέρους. Ίσως να αποσαφηνίσουμε ότι η χρηματοδότηση της σύμβασης τρίτου μέρους θα πρέπει να αποκαλυφθεί μόνο στο δικαστή και όχι στον καθού, γιατί Φυσικά η σύμβαση αυτή θα περιλαμβάνει όλη τη στρατηγική της ε, διαφοράς. Ό,τι αφορά τώρα το πεδίο εφαρμογή. Θα έλεγα ότι κάποια σημαντικά νομοθετήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προσθεθούν στο παράρτημα, δηλαδή χάρη στον τομέα του ανταγωνισμού για να καλύψουν αυτό που έχουμε τουλάχιστον στο Βέλγιο τώρα και για τον ορισμό της ζημίας θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι θα πρέπει να μιλάμε για οικονομική ζημία ή ηθική ζημία, ηθική βλάβη. Είναι το χάρη την προστασία των δεδομένων στο σκάνδαλο με το Facebook. Κατόπιν, σε σχέση με την ενημέρωση των καταναλωτών, υπάρχουν κάποιες διατάξεις στην πρόταση που υποχρεώνουν τον έμπορο να καλύψει το κόστος της ενημέρωσης των καταναλωτών. Το υποστηρίζουμε αυτό και προτείνουμε περαιτέρω ο νομοποιούμενος φορέας να εγκρίνει το περιεχόμενο των πληροφοριών που δίνονται από τον έμπορο στον καταναλωτή. Έχουμε ένα παράδειγμα Ο ε, πάροχος τηλεπικοινωνίας, ε, στον οποίο σκίσαμε μήνυση, διτέχθηκε από το δικαστήριο να ενημερώσει τους καταναλωτές του για την ε, ύπαρξη ε, Συλλογική αγωγή εναντίον του και έστειλε μια εντελώς παραπλανητική επιστολή. Έτσι λοιπόν οι πληροφορίες που δόθηκαν από τον ε, έμπορο πρέπει να ελέγχονται είτε από τον υπουργμένο είτε από το δικαστή. Και όπως ήδη υπόθηκε χρειάζεται και αποσαφήνιση σε σχέση με το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Ποιοι κανόνες θα ισχύουν δηλαδή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν μακρηγόρησα, οπότε μην διστάσετε να θέσετε ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τους δύο τελευταίους ομιλητές για την παρουσίασή τους. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε ερωτήσεις. Θέλετε το λόγο? Κύριος Φάλκεν. Yeah, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις ε, πολύ χρήσιμες ε, παρουσιάσεις. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είχα ρωτήσει και νωρίτερα, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. Προς ε, εσάς λοιπόν ρωτώ εάν θεωρείτε ότι η πρόταση με κάποια τροποποίηση της μπορούσε να οδηγήσει σε μια βιομηχανία των αγωγών, αν φοβάστε μια τέτοια εξέλιξη. Και αυτό το λέω γιατί όταν ε, βλέπουμε όλες αυτές τις ε, λεπτομέρειες που προβλέπονται, βεβαίως μπορεί να φαίνονται πολύ λεπτομέρειες, αλλά ταυτόχρονα σε, αυτό, σε αυτή τη φούσκα που λέγεται Βρυξέλλες, βλέπουμε πολύ συχνά ότι προτείνονται λύσεις οι οποίες ε, αποβαίνουν σ' μιας βιομηχανίας των αγωγών και τελικά δεν ασχολείται κανείς με τις λεπτομέρειες. Θεωρείτε λοιπόν ότι η επέκταση σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα θα μπορούσε να αποτελέσει μια επικίνδυνη εξέλιξη στον χώρο της δημόσιας υγείας, στον χώρο του, χώρο του περιβάλλοντος, κάτι τέτοιο θα ήταν οπωσδήποτε πολύ χρήσιμο και γι' αυτό θα ήθελα και τις δικές σας εκτιμήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προς τον κύριο Ναβάμ και την ε, συναδελφό του απευθύνομαι κυρίως με την ερώτησή μου και χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω την ε, αναγκαιότητα για ενισχυμένη προστασία των καταναλωτών για το θέμα αυτό και ως συγκεκριτής δεν μπορώ παρά να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι λαμβάνεται υπόψη αυτή η ανάγκη προστασίας ε, ταυτόχρονα ωστόσο γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και κίνδυνοι καταχρήσεων. Με το παράδειγμα λοιπόν ε, της υπόθεσης αυτής που έχουμε και της νομοθεσίας που έχουμε στο Βέλγιο, θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχει προβλέψει η βελγική νομοθεσία κινδύνους που οπωσδήποτε θα έχουν το μεταξύ εντοπιστεί. Και για να δώσω το παράδειγμα της Thomas Cook, θα μπορούσαν να οδηγήσουν παραδείγματι στο να ε, καθοδηγήσει ε, πίσω από τα παρασκήνια κάποιος ανταγωνιστής της εταιρείας μια συλλογική αγωγή κατά του αντιπάλου του, του εμπορικού. Η προστασία του καταναλωτή, την οποία συμμερίζουμε τους, δεν θα μπορούσε να οδηγήσει και σε παρεκτροπές και αν ναι, και πιστεύω ότι το μέλημα μας απασχολεί όλους η βελγική νομοθεσία έχει ορίσει διασφαλιστικές δικλείδες. Και αν όχι, θεωρείτε ότι θα ήταν σκόπιμο να υπάρχουν τέτοιες διασφαλιστικές δικλίδες. Κύριος Φώσης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μια σειρά από ερωτήσεις με απασχολούν. Η πρώτη έχει να κάνει με το λεγόμενο forum shopping που στο πρώτο τμήμα κυρίως ακούσαμε περισσότερο, στο δεύτερο λιγότερο εθίγη. Ξέρω ότι δεν ήταν και αντικείμενο των παρουσιάσεων τόσο, αλλά θα ήθελα να έχω μια εκτίμηση. Μια μελέτη παραδείγματι της Επιτροπής έδειχνε ότι υπάρχει κίνδυνος για forum shopping, δηλαδή επιλογή της πιο ευνοϊκής δικαιοδοσίας ε, ότι, και μάλλον ότι θέλει να ενημερώνει αυτή η μελέτη για, την, για τον κίνδυνο. Και επομένω, πώ μπορούμε να αποφύγουμε μια τέτοια ε, εναλλαγή ε, και αναζήτηση της πιο ευνοϊκής, της πιο απλής ενδεχομένως, εν πάση της πιο αποδοτικής δικαιοδοσίας και πώς μπορεί να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος. Θα ήθελα και οι τελευταίοι ομιλητέ μα να αναλύσουν αυτόν τον κίνδυνο για αναζήτηση πιο ευνοϊκή δικαιοδοσία και κυρίως τις παραμεθόριες περιοχέ σε περίπτωση των ε, συλλογικών αγωγών που βλέπω ότι θα ήταν πιο μεγάλο ο κίνδυνο ή γενικώ αν τον κρίνει τον κίνδυνο αυτό υψηλό ή μη και αν θεωρούν ότι ο κανονισμός Βρυξέλλες 1α ή ε, Ρώμη 1 χρειάζονται τροποποίηση. Επίσης, για να συμφωνήσω και με, για να συνεχίσω μάλλον στην ερώτηση του κύριου Βέλκεν, για το, βιομηχανία αυτή, η φάμπρικα των ε, ε, αγωγών. Ξέρω ότι μια τέτοια ερώτηση δεν έχει νόημα, δεν έχει σαν επιδίωξη να κλείσει το θέμα. Απλώς ξέρω ότι δεν περιορίζονται στο να πούν οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες ότι τους ικανοποιεί και μόνο να ε, ικανοποιείται το δικαίωμα του καταναλωτή. Και θα ήθελα να πάω λίγο παραπέρα την ερώτηση λοιπόν για να πω ότι με τις εξελίξεις που βλέπουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στις ε, κάτω χώρες είναι ο κίνδυνο υπαρκτό και για όλου, δηλαδή τα κριτήρια που μπορεί να απορρέουν από την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επαρκώ προσδορισμένα ώστε να αποφευχθεί να αποτραπεί ένα τέτοιο κίνδυνο. Ή μήπω. ο αποκλεισμός της ε, εργολαβικής αμοιβή για τους ε, δικηγόρους σε περίπτωση μόνο δηλαδή ε, δικαίωσης θα ήταν μια λύση για το μοντέλο opt-out επίσης. Θα ήταν σκόπιμο να φέρετε στις περιπτώσεις αυτές. Αλλά ο ενάγων μπορεί να έχει αντίληψη του ότι είναι μέρος μιας τέτοιας συλλογική αγωγής, μιας τέτοιας διαδικασίας και να κάνει το opt-out, να επιλέξει δηλαδή να μην συμπεριληφθεί. Μπορεί, υπάρχει η δυνάμει αυτή η αντίληψη, έχει κάποιο νόημα αυτό το opt-out. Όσο και αν μου φαίνεται σκόπιμο, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Θα έχουμε δηλαδή κάποια στιγμή προκαταρκτικά ενδεχομένως της ε, εκκίνησης της αγωγής, ε, το πώς είναι οι ενδιαφερόμενοι, γιατί όγκο αποζημιώσεων μιλούμε κτλ. Και μια άλλη, ένα άλλο θέμα που πάλι έχει να κάνει με τις δυνατότητες για την πρακτική εφαρμογή στον χώρο του περιβάλλοντος που ανέφερε και ο συνάδελφος Βούλκερ. Πολύ ωραίο ακούγεται, αλλά αν φερειπίνω εγώ ρηπάνω ε, τον ατμοσφαιρικό αέρα Πώς είναι δυνατόν να προσδοριστεί ε, ποιο ζημιώνεται από αυτό. Ας πούμε ότι έγινε, ότι η ρήπανση προκύπτει, η γεννάτε στο ε, Αμβούργο, αλλά φτάνει το, ο ρήπος μέχρι το Μόναχο. Πού θα ορίσω ε, το πεδίο συνεπειών, πού θα τραβήξω τη γραμμή. Και επίσης, επειδή υπάρχει σχετική αν η αντίστοιχη ρήτρα στο άρθρο 80 του κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Βλέπω ότι θα ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί να το όρια στην υπόθεση αυτή και στον τομέα των θεμελιωδών ελευθεριών ε, δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να προεξοφλούμε ότι κάποιος μπορεί να διεκδικήσει ένα τόσο ε, ή ότι οφείλει να διεκδικήσει ένα τόσο προσωπικό δικαίωμα ας πούμε με την υπόθεση Facebook, Cambridge Analytica ή ενδεχόμενο hacking προσωπικών δεδομένων που μπορεί να προκύπτει η πετιότητα κάποιες επιχείρησης. Πώς θα κριθεί το ποιος τελικά επλήγει από την παραβίαση αυτή ή από την ε, υπετιότητα. Ε, όταν έχουμε να κάνουμε με ένα δικαίωμα θεμελιώδες και το και το οποίο δικαίωμα θεμελιώδε δεν μπορεί κανεί να ασκήσει. Τουλάχιστον δεν μπορώ εγώ να θεωρήσω ότι κάποιο θα το ασκήσει στο όνομά μου. Μήπω θα ήταν καλύτερο να ξεχάσουμε το opt-out, αλλά να έχουμε ένα πιο συνειδητό opt-in. Συγγνώμη που με μακρηγόρησα. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω. Ήλπιζα μάλλον οι ερωτήσει να μην είναι τόσο μεγάλε, να, οι απαντήσει να είναι μεγαλύτερε. αλλά έχουμε 14 λεπτά, θα προσπαθήσουμε να μείνουμε εντό χρόνου. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τους προσκεκλημένους να επιλέξει ο καθένας να απαντήσει στις ερωτήσεις που τον αφορούν ή την αφορούν. Ο κύριος Σόλτ έχει στήσει να παρέμβει. Ναι, ευχαριστώ. Έχουμε τον ε, Ραφαλ Μερό που θέλει να απαντήσει στον ε, κίνδυνο καταχρήσεων. Έχει συμμετέχει και στη δική μας μελέτη. Ο κίνδυνος καταχρήσεων ε, είναι κάτι που επιβάλλεται όταν συζητάμε για συλλογικές αγωγές. Θέλω να κάνω δύο σύντομες παρατηρήσεις για να απαντήσω στους κυρίους Βαλκαν και Ντιντιέ. Η εμπειρία μας στη Γαλλία μέχρι τώρα είναι το αντίθετο. Οι συλλογικές αγωγές δεν λειτουργούν καθόλου. Δεν υπάρχει καν κατάχρηση. Και αν αναρωτηθείτε, οι κύριε ενώσει καταναλωτών στη Γαλλία που μπορούν να προβούν σε συλλογικέ αγωγέ θα σα πούνε ότι δεν θέλουν πια, γιατί είναι ανίκανος, ε, ανίκανες ε, να ε, προσφύγουν στη δικαιοσύνη επειδή είναι πάρα πολύ βαριές αυτές οι διαδικασίες. Επομένως έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα από την κατάχρηση. Επίσης προβλέπονται κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες στο κείμενο και στην έκθεση που σας υποβάλαμε που μπορούν να απομακρύνουν αυτόν τον κίνδυνο κατάχρησης. Τρίτη παρατήρηση κύριος Βόλκεν μιλούσε για μια βιομηχανία αγωγών. Μάλλον η απουσία του ευρωπαϊκού κειμένου ευνοεί ε, κάτι τέτοιο και στην Ευρώπη, κυρίως ε, σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό και τις αγωγές για θέματα ανταγωνιστού, έχετε, παραδείγματο χάρη, κάποια δικηγορικά γραφεία ήδη που κάνουν forum shopping, επιλέγουν την καλύτερη δικαιοδοσία ακριβώ γιατί δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεν υπάρχουν ασφαλιστικέ δικλείδε για να αποφευθούν αυτέ οι καταχρήσει. Στον τομέα τη κατανάλωση, ε, μια κατάχρηση ε, είναι σίγουρα ε, η περίπτωση ότι όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει καμία εμπειρική μελέτη που μας δείξει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν τέτοιες καταχρήσεις. Έχουμε πολλές φορές ψευδείς ειδήσει για το καταναλωτικό τομέα. Σε ό,τι αφορά όμως τον ανταγωνισμό που κινείται το χρήμα, η έλλειψη νομοθεσίας δημιουργεί τις καταχρήσεις. Δεύτερη παρατήρηση και θα σταματήσω. Προσπαθήσαμε στην έκθεση της Trans Europe να περασπίσουμε τον εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών. Μάλιστα προτείναμε να καταστούν υποχρεωτικές. Θέλαμε και εδώ να ευχαριστήσουμε την προσοχή σας, αλλά για να είναι αποτελεσματική αυτή η τρόπη θα πρέπει να είναι, αποτελεσματική και, ε, να είναι αποτελεσματικές και οι διαδικασίες στο δικαστήριο. Δηλαδή κανένας δεν θα κάτσει στο διαπραγματευτικό τραπέζι αν δεν φοβάται ότι θα καταδικαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης του κράτους. Αν θέλουμε εναλλακτική τρόπο επίλυσης διαφορών να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει και τα δικαστήρια να είναι αποτελεσματικά. Έτσι λοιπόν, έτσι θα φτάσουμε να λύνουμε τα θέματα με ένα φιλικό τρόπο, με διαπραγμάτευση ε, και έτσι ώστε να μην επιβαρύνουμε και τα κρατικά δικαστήρια. Θα πρέπει όμως το κείμενο να είναι και στο ύψος των περιστάσεων. Σας ευχαριστώ. Η καθηγήτρια Augenhofer. Um, um Λοιπόν, δεν φοβάμαι τον ενδεχόμενο καταχρήσεων να εγκριθεί η πρόταση. Αυτό που φοβάμαι, μάλλον, είναι ότι ε, κάποια από τα άρθρα δεν είναι αρκετά φιλόδοξα. Δεν βλέπω, λοιπόν, πιθανότητα καταχρήσεων και όπως είπε και ο συνάδελφος δεν υπάρχουν εμπειρικές μελέτες σχετικά με το πώς έχει γίνει κατάχρηση και πόση κατάχρηση έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του συστήματος. Δεν έχει παρατηρηθεί κατάχρηση στην υπόθεση της Volkswagen στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχε επιτροπή εξεταστική και οι καταναλωτές ε, ρωτήθηκαν αν προτιμούν χρηματική αποζημίωση ή επισκευή του αυτοκινήτου και ε, πήραν ένα ποσό κατά αποκοπή. Γι' αυτό λοιπόν αυτό δεν καθιστά κατάχρηση. Μάλιστα, αν δείτε και τις δηλώσεις τύπου της Volkswagen στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα νομίζετε πως οι δηλώσεις προέρχονται από δύο διαφορετικές εταιρείε. Γιατί στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, η δήλωση κάπως ε, έλεγε ότι «Ω, σας παρακαλούμε, δεν το ξανακάνουμε, μη σταματάτε να αγοράζετε τα αυτοκίνητα», ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε ότι οι καταναλωτές δεν θα πάρουν δεκάρα από εμά. Υπάρχει λοιπόν διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Τώρα, περιπτώσεις κατάχρησης λόγω της αναζήτησης ευνοϊκής δικαιοδοσίας στις αρχές του έτους ακούσαμε ότι αν οι καταναλωτές ασκήσουν αγωγή και αν ε, η αγωγή ασκηθεί από μια εγκεκριμένη οντότητα σε άλλο κράτος μέλος, τότε οι καταναλωτές ε, χάνουν τα δικαιώματά τους στο... στη χώρα τους. Οι εγκεκριμένε οντότητε λοιπόν είναι προβληματικέ εκτό αν αλλάξει ο αντίστοιχο κανονισμό. Πρέπει η αγωγή να υποβάλλεται στο, στην έδρα του αναγόμενου. Δεν ξέρω λοιπόν πώς με αυτόν τον τρόπο ε, θα γίνει αυτή η αναζήτηση ευνοϊκής δικαιοδοσίας, αυτό το forum shopping. Υπάρχει λοιπόν αυτή η απόφαση από τον Ιανουάριο του 2018 που ε, ξεκαθαρίζει το τοπίο, όμως τώρα θα δώσω το λόγο στην συνάδελφο για την ερώτηση και θα επιστρέψω. Ναι, θα ήθελα να δώσω την απάντηση τώρα, αν μου επιτρέπετε. Στην ερώτησή σας. Υπάρχει κίνδυνος ε, να υποκινεί από τα παρασκήνια ένας ανταγωνιστής μια τέτοια ε, αγωγή. Δεν νομίζω. Γιατί η οντότητα που πρέπει να ξεκινήσει αυτή την αγωγή στο Βέλγιο πρέπει να είναι μέλο τη σχετική οργάνωση ε, Ένωση Συμβουλίου του Βελγίου ή να έχει εγκριθεί από το Υπουργείο και πρέπει να έχει νομική προσωπικότητα από τριετία τουλάχιστον. Άρα ο, ο έλεγχο είναι πραγματικό. Δεν μπορεί κανεί να ιδρύσει μια ένωση ad hoc για να αναλάβει μια συγκεκριμένη συλλογική αγωγή. Και επίση στην ερώτηση αν θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει σε μια φάμπρικα των ε, αγωγών. Θα σας απαντήσω πολύ πρακτικά. Στο Βέλγιο που υπάρχει ο νόμος αυτός εδώ και τέσσερα χρόνια είμαστε η μόνη εντότητα που έχει εκκινήσει αγωγές συλλογικές και συνολικά από το 2014 έχουμε καταθέσει 7 αγωγές. Επομένως δεν υπάρχουν καταρχάς πολλά κίνητρα για να ξεκινήσει κανείς γιατί είναι περιορισμένο το ε, οικονομικό κέρδος. Εμείς δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα, το κάνουμε μόνο προς το συμφέρον του καταναλωτή ως Ένωση ε, Δικαιωμάτων των Καταναλωτών. Ε, όχι μόνο δεν κερδίζουμε, μάλλον μπαίνουμε μέσα οικονομικά. Γι' αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε και τις προτάσεις μας για να βελτιωθεί το οικονομικό σκέλος, γιατί για μας είναι πολύ δύσκολο. Άρα λοιπόν φάμπρικα αγωγών δεν βλέπω αν δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο θα μπορούσε να προκύψει. Ναι, ευχαριστώ. Θα απαντήσω στην ερώτησή σας για το opt-out ε, ως ε, επιλογή καταρχήν. Ε, ίσως θα μπορούσε να είναι καλύτερη η λύση του opt-in εάν είναι δύσκολο να υπολογιστεί ο όγκος της ζημίας ο αριθμός των καταναλωτών, αλλά εμείς βλέπουμε από την εμπειρία μας ότι είναι ευχερής ο προσδιορισμός του αριθμού των καταναλωτών. Στην περίπτωση του Μασκού είχαμε 220 περίπου επιβάτες της, ε, της συγκεκριμένης της συγκεκριμένης εταιρείας. Ήταν εύκολο να εντοπιστούν και άρα να προκύψει το, η επιλογή του opt-out ε, εύκολα. Είχαμε μια άλλη ε, αγωγή για συμβάσεις αγοράς, Pampers που δεν παραδόθηκαν ποτέ από την Αμερικανική εταιρεία εκπτωτικών πωλήσεων, γκρουπών. Και πάλι αυτοί ήξεραν πολύ καλά με ποιον είχαν συνάψει τη σχετική σύμβαση πώληση. Επομένω, ήταν πολύ πιο χρήσιμο το opt-out. Στην υπόθεση πρόξιμου τη εταιρεία τηλεπικοινωνιών που ανέφερα νωρίτερα, Ακριβώ η πρόξιμο ήξερε πολύ καλά ε, πόσους καταναλωτές ε, αφορούσε η σχετική ενημέρωση. Μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του είτε με το email είτε με το τηλέφωνο Υπάρχουν περιπτώσει βέβαια είναι, όπου είναι δύσκολο ο υπολογισμό των καταναλωτών, οπότε ενδεχομένω το opt να φαινόταν πιο χρήσιμο. Η πιο σωστή λύση. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Α, η κυρία Άγκουνχόφερ. Ναι, αν μου επιτρέπετε μια ερώτηση, μάλλον δύο ερωτήσεις που δεν έχουν ακόμη απαντηθεί, δεν ξέρω αν έχουμε ακόμα χρόνο για το περιβάλλον. Περιβαλλοντική προστασία και χωρίς να ισχυρίζομαι ότι είμαι ειδική στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος. Ε, το πράγμα που δώσατε, Αμβούργο και Μόναχο, Βερολίνο, τέλο πάντων ένα εργοστάσιο στο Αμβούργο ε, έχει ρηπογόνο δραστηριότητα η οποία φέρνει αποτελέσματα και στο Βερολίνο. Δεν υπάρχει ζήτημα, δεν υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με την παραβίαση των περιελωτικών κανόνων, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και επίσης το άρθρο 80 του κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επισημάνατε είναι μια διάταξη μάλλον απογοητευτική ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, γιατί προβλέπεται ως επιλογή μόνο προαιρετική για τα κράτη-μέλη δηλαδή, να έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει ένα κράτος το αν μια ένωση καταναλωτών θα αναλάβει τη δυνατότητα για αγωγή. Και αυτό λέω ότι είναι απογοητευτική, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτική αυτή η κλίση. και θεωρώ ότι αν τελικά εγκριθεί η πρόταση ε, για μένα δεν θα είναι πρόβλημα το ότι υπάρχει επικάλυψη, δεν βλέπω εγώ πρόβλημα επικάλυψης δηλαδή μεταξύ των διατάξεων του αντίον. θα είναι πρόοδο η εισαγωγή αυτή τη πρόταση στο νομοθετικό πλαίσιο γιατί η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι επαρκή. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, σε σχέση με το Forum Shopping, δύο σχόλια. Καταρχήν, όσο δεν έχουμε ένα αρμονισμένο μέσο, όντω υπάρχει ένα τέτοιο κίνδυνο και είναι όλο ένα και πιο αυξημένο. Και ακριβώ ε, πρέπει να έχουμε ένα εναρμονισμένο μέσο που να περιορίζει τον κίνδυνο του forum shopping. Δεύτερο, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά σε σχέση με την άγρια δικαιοδοσία, ακόμη και με εναρμονισμένου κανόνε. Γιατί, αν ρωτήσετε του ε, κύριου πρωταγωνιστέ στον τομέα του ανταγωνισμού που προβαίνουν ήδη σε forum shopping, η επιλογή τους ε, στο να πάνε στη μικρή και όχι σε άλλα εξαρτάται από τα αγγλικά παραδείγματο χάρη. Υπάρχει ένα forum shopping προς ε, το δικαστήριο των κάτω ε, γιατί γίνεται η διαδικασία στα αγγλικά. Και επομένως αυτός είναι ένας από τους παράγοντες που ε, οθεί τις υποθέσεις ε, προς ε, την Ολλανδία. Το ίδιο συμβαίνει και με την Αγγλία. Υπάρχουν κάποια δικηγαρικά γραφεία αγγλοσεξιονικά που μιλούν αγγλικά και χειρίζονται καλύτερα τη γλώσσα. Έτσι λοιπόν αν είχαμε ένα αρμονισμένο σύστημα ίσως θα όταν κάπως αυτός ο κίνδυνος αλλά δεν θα εξαλειφόταν ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους μας που μοιράστηκαν τις γνώσεις τους μαζί μας σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το επόμενο σημείο είναι και κλεισμένο το θυρών, έτσι λοιπόν πρέπει να ζητήσω από όλους ε, όσους δεν ε, έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται εδώ να αποχωρήσουν.